Okay, um, Καλημέρα. Καλώς ήρθατε. Περνάμε σημείο 9 της ημερησίας διάταξης και με ιδιαίτερη χαρά καλωσορίζω το τον Γενικό Γραμματέα του ΟΣΑ, τον κύριο Αγχέλ Γκουρία. Δεύτερη φορά έρχεται ε, σε συνεδρίαση της Επιτροπής μας και σας ευχαριστώ ιδιαίτερα. Είμαι σίγουρη πως θα έχουμε μια ενδιαφέρουσα ανταλλαγή απόψεων. Υπάρχουν διάφορα ενδιαφέροντα έγγραφα, τα οποία εγώ τα φόρτωσα στους βοηθούς μου για να μπορέσω να διαβάσω τα επίσημα έγγραφα, εκθέσεις και τέτοια πράγματα και είμαι σίγουροι πως ε, θα τα συζητήσουμε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης. Να σας δώσω λοιπόν το λόγο να κάνετε κάποια αρχικά σχόλια και μετά θα περάσουμε σε ερωτοαπαντήσεις για να περιοριστούμε σε πεντάλεπτα ερωταποκρίσεων. Ελπίζω δηλαδή να επικρατήσει η πειθαρχία. Λοιπόν, Ανχέλ, έχετε τον λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Η γραμματεία πρέπει να έχει ήδη μοιράσει κάποια έγγραφα. γενικές πληροφορίες για την παγκόσμια οικονομία. Θα αναφέρω τα κυρία σημεία, μετά θα αναφερθώ στην ευρωπαϊκή οικονομία. Πρώτα απ' όλα η κρίση ε, υπάρχει ακόμα και μας έχει αφήσει τέσσερα σημεία σκληρονομιά. Πρώτον η χαμηλή ανάπτυξη. Η παγκόσμια ανάπτυξη είναι κάτω από το 3% η χαμηλότερη δηλαδή εδώ και αρκετά χρόνια. Αναμέναμε να φτάσουμε έτσι το, το ρελαντί το 4% αλλά είμαστε αρκετά κάτω από αυτό λόγω της κρίσης. Στις είπα παρά το κλείσιμο του δημοσίου η ανάπτυξη έρχεται και παρόλες τους πολιτικούς καυγάδες και τις αυτόματες περικοπές, κάτι το οποίο δείχνει πόσο δυναμική είναι αυτή η οικονομία. Χωρίς ε, τις αυτόματες περικοπές ε, των δαπανών, θα είχαν 1-1,5% ε, παραπάνω ανάπτυξη, είπα. Οπότε προχωράνε, αλλά ταυτόχρονα λόγω των αυτομάτων ε, περικοπών μειώνουν ε, πάρα πολύ γρήγορα το έλλειμμα. Κάτω από το 4% είναι τώρα. Οπότε θα ανακάμψουν γρηγορότερα αργότερα. Στην Ιαπωνία η ανάπτυξη αναμένεται να επιβραδυνθεί του χρόνου γιατί τα δημοσιονομικά κίνητρα πλέον δεν θα υπάρχουν και βεβαίως ο λόγος είναι πως η Ιαπωνία έχει 220-230% του ΑΕΠ χρέος. Οπότε έχουν χαλαρή νομισματική πολιτική, αλλά δεν μπορούν να συνεχίσουν να έχουν τα ίδια δημοσιονομικά κίντρα. Και επίσης ε, έχουν έναν ε, πληθωρισμό 2%. Φανταστείτε να έχουν 2% πληθωρισμό και χρέος 250% του ΑΕΠ. Πολλαπλασιάστε το, το 250 επί 2%. Ας υποθέσουμε τα πραγματικά επιτόκια είναι 2%. Οπότε πρέπει να έχουν 5% ανάπτυξη κάθε χρόνια να πληρώνουν τους τόκους. Έτσι, πρέπει να έχουν ε, πλεόνασμα, με συγχωρείτε, 5% κάθε χρόνο για να πληρώνουν τους τόκους. Έχουν λοιπόν ένα έλλειμμα ε, διψήφιο, οπότε ο μετασχηματισμός που χρειάζεται είναι τεράστιος. Τώρα, στην Ευρώπη ε, δεν είναι μεγάλη ανάκαμψη, είναι και άνηση, υπάρχει μια μικρή ανάπτυξη στις περισσότερες χώρες εκτός της Ευρωζώνης, αλλά στην Ευρωζώνη έχουμε ύφεση για δεύτερο χρόνο, εμείς λέμε μείον 0,4% και λίγη βελτίωση βραχυπρόθεσμα, λέμε 1% του χρόνου και 1,6% το 2015. Τίποτα το σπουδαίο δηλαδή. Δυστυχώς. Αυτή είναι η πρώτη κληρονομιά της ε, κρίσης. Η δεύτερη, η ε, υψηλή ανεργία. Τα νούμερα τα ξέρετε, αλλά είναι απαράδεκτα υψηλά. Στον ΩΣΑ κατά μέσο όρο 8% ανεργία, 16% ανεργία των νέων. Αυτός είναι ο μέσος όρος. Στην Ευρωζώνη 12% ανεργία και αυξάνεται και η ανεργία των νέων 25-30% σε χώρες όπως η Ισπανία, η Ιταλία, 35% και μετά Ελλάδα, μιλάμε για 50-55%. Οπότε υψηλή ανεργία διπλή και τρίδιπλή ανεργία των νέων και ένα τέταρτο στοιχείο που είναι αυτοί οι οποίοι δεν είναι σε, ε, ούτε απασχολούμενοι ούτε στην εκπαίδευση ούτε οτιδήποτε άλλο. Τέσσερα άσχημα στοιχεία όσον αφορά την απασχόληση. Ποια είναι η τρίτη κληρονομιά που μας άφησε η κρίση. Είναι η εισοδηματική ανισότητα η οποία αυξάνεται. Τι εννοούμε ανισότητα εισοδήματος πόσες φορές το εισόδημα του χαμηλότερου 10% ε, είναι το εισόδημα του ανώτερου 10%. Εννέα φορές. Και λοιπόν, τι έγινε. Ε, να σας πω τι έγινε. Πριν από μία γενιά ήταν 6 φορές μεγαλύτερο το, το εισόδημα, η διαφορά αυτή. Οπότε αυξήθηκε η εισοδηματική ανισότητα αυξανόταν αλλά οξύνθηκε. Στη ΣΥΠΑ είναι 14%, στο Μεξικό είναι 25 φορές, ε, στη Βραζιλία είναι 50 φορές το πολλαπλάσιο αυτό και όπως σας είπα τα πράγματα επιδεινώνονται. Και πρακτικά καμία χώρα δεν εξαιρείται. Χαμηλή ανάπτυξη λοιπόν, υψηλή ανεργία, ανισότητες και τέταρτον η κοινή γνώμη χάνει την εμπιστοσύνη της ε, στο κράτος. Εμείς μόλις δημοσιεύσαμε μία σχετική έκθεση, μία λέγεται το κράτος με μία ματιά και η άλλη... λέγεται πώς έχει η ζωή. Βλέπουμε λοιπόν μία μείωση στην εμπιστοσύνη του κοινού. Εμπιστοσύνη σε τι, στα πάντα. Σε προέδρους, πρωθυπουργούς, ε, σε κόμματα, στις πολυεθνικές, ε, στις τράπεζες, στα κοινοβούλια, σε διεθνείς οργανισμούς. Ό,τι οικοδομήσαμε τα τελευταία 100 χρόνια ε, πλέον δεν το εμπιστεύεται ο κόσμος, είναι κοινικός. Δεν θεωρούν πως μπορούμε να λύσουμε τα προβλήματα. Αυτό συμβαίνει. Αυτό είναι το πλαίσιο. Λοιπόν, αυτά μας άφησε η κρίση. Ποια είναι η διάγνωση λοιπόν της σημερινής οικονομίας. Κοιτάξτε, οι Αμερικανοί λένε πως ε, δουλεύει στο full είναι μία, μία έκφραση. Αυτοί λένε ότι δουλεύουν και οι τέσσερις κύλινδροι. Κανένας λοιπόν δεν δουλεύει θα έλεγα η οικονομία και στους τέσσερις ε, κυλίνδρους. Ποιοι είναι αυτοί οι τέσσερις κυλίνδροι? Είναι εμπόριο, επενδύσεις, οι ε, BRICS, και η ανάπτυξη. Λοιπόν, οι BRICS ε, είναι γύρω στο 4-5% η ανάπτυξη, έχουν προβλήματα με τις διαπραγματεύσεις, δεν μπορούν καν να διευκολύνουν το ε, διασυνοριακό εμπόριο, πόσο μάλλον για έναν επόμενο γύρο παγκοσμίου εμπορίου. Οπότε είναι πάρα πολύ δύσκολο να μιλήσουμε για διατλαντική συμφωνία που θα είναι πάρα πολύ σημαντική. Αν τα καταφέρουμε στο καλό θα είναι, αλλά είναι ο εύκολο στόχο. Αν δεν τα καταφέρουμε ούτε εκεί, θα είναι απογοητευτικά τα πράγματα. Δεν έχουμε λοιπόν το εμπόριο ω ατμομηχανή όπως ήταν παλιά. Δεύτερον, επενδύσει. Οι επενδύσει αυξάνονται με 1,7%. Θα έπρεπε να αυξάνονται με 3-4%. Η ΕΠΑ είναι στο 1,5%. Χαμηλό, ιστορικό χαμηλό. Γιατί έχει σημασία αυτό, γιατί οι επενδύσει είναι η αυριανή ανάπτυξη και δεν συμβαίνουν, δεν υπάρχουν. Οπότε, άλλο στοιχείο, πίστοση, η πίστη. Δηλαδή η ανάκαμψη του χρηματοπιστωτικού συστήματος και το ότι οι τράπεζες δεν φτάνει μόνο να επιζήσουν και να ανακεφαλαιοποιηθούν και να έχουμε μία εποπτική αρχή, ε, πρέπει να δανείζουν κιόλας πρέπει να δανείζουν και δεν δανείζουν. Η μέση αύξηση της πίστης στον ΩΣΑ είναι 0, που βεβαίως σαν κάθε μέσος όρος υποκρύπτει το ότι αυξάνεται στις ΗΠΑ και στην Ιαπωνία και είναι αρνητική στην Ευρωζώνη, μείον 4% για να είμαι ακριβής. Οπότε, δεν υπάρχει καμία έκπληξη βεβαίως. Και τέλος η BRICS που ήταν επίσης ατμομηχανή και τώρα επιβραδύνουν. Οπότε δεν λειτουργούν, θα έλεγα, αυτοί οι τέσσερις κύλινδροι του κινητήρα όπως θα μπορούσαν, οπότε τι πρέπει να κάνουμε. Πρέπει να έχουμε μια προσέγγιση πάλι τετραπλή, δηλαδή διαρθρωτικές πολιτικές, κοινωνικές, για τους πιο αδύναμους, πράσινη ανάπτυξη, γιατί υπάρχει πρόβλημα με τη φύση και θα πέσουμε στον τοίχο και τέταρτον θεσμικά ζητήματα. Οπότε βασικά Τι σημαίνει διαρθρωτικές αλλαγές. Θα λέμε συνέχεια τι σημαίνει αυτό. Τα παλιά κλασικά. Εκπαίδευση, καινοτομία, ανταγωνισμός, φορολογικό σύστημα, σύστημα υγείας, ευελιξία στην αγορά εργασίας, ευελιξία στην αγορά προϊόντων, η σχέση μεταξύ ερευνητικών κέντρων και πανεπιστημίων και ιδιωτικού τομέα και αγοράς, αποκέντρωση, πώς θα χρηματοδοτηθούν οι υποδομές, αυτά εννοούμε διαρθρωτικά. Και σημαίνει το πώς θα συνεχίσουμε να παρέχουμε δεξιότητες που απαιτούνται για να είναι κανείς ανταγωνιστικός. Μετρήσαμε μετά από τρία χρόνια δουλειάς κάναμε την πρώτη σύγκριση δεξιοτήτων. Είναι κάτι διαφορετικό από το έγγραφο που βγάζουμε για την πίζα που αφορά τους 15χρονους μαθητές και θα βγει αυτή η έκθεση στις 3 Δεκεμβρίου. Συγκρίνουμε 70 χώρες για, για τα αποτελέσματα της εκπαίδευσης. Εδώ πέρα μιλάμε για τους ενηλίκους, αν έχουν τις κατάλληλες δεξιότητες στη δουλειά τους. Και επιστώσαμε ενδιαφέροντα πράγματα. Η Κορέα, παραδείγματος χάρη, έχει τις χειρότερες ε, γενιές που φεύγουν από την αγορά εργασία και τις καλύτερες που μπαίνουν στην αγορά εργασία και χώρε όπως το Ηνωμένο Βασίλειο ή ΙΠΑ καμία ορατή διαφορά μεταξύ των γενεών που φεύγουν και αυτών που μπαίνουν στην αγορά εργασίας. Δηλαδή δεν υπάρχει βελτίωση. Η Ισπανία δεν τα πήγε πάρα πολύ καλά. Οπότε το ερώτημα είναι το εξής. Το θέμα δεν αφορά τα διπλώματα και τα πτυχία. Αφορά τις δεξιότητες που χρειάζεται κανείς για να κάνει τη δουλειά του. Είναι κρίσιμη λοιπόν η κατάσταση. Αυτά είναι τα διαρθρωτικά. Τα κοινωνικά γιατί όσο σφιχτή και αν είναι οι προπολογισμοί, πάντα πρέπει να υπάρχει περιθώριο προστασίας των αδυνάμων, γιατί υπάρχουν πολλά εκατομμύρια θύματα της κρίσης. Στον ίδιο τον όσα υπάρχουν 48 εκατομμύρια άνεργοι και το πρόβλημα είναι πως είναι 15 εκατομμύρια παραπάνω από όσους υπήρχαν πριν την κρίση. Ακόμα και με την ανάπτυξη της ΕΠΑ έχουμε 15 εκατομμύρια περισσότερους άνεργους. Τώρα, Τέλος. Για το τραπεζικό σύστημα της Ευρώπης και μετά θα περάσουμε στις ερωτήσεις και απαντήσεις και κάτι για τους φόρους. Το τραπεζικό σύστημα γενικώ ανακάμπτει, έχει βελτιωθεί η κατάστασή του γιατί ε, εκεί πέρα προέκυψε το πρόβλημα από τη ΣΥΠΑ, Ευρώπη και μετά εξαπλώθηκε σε όλο τον κόσμο. Το θέμα είναι ότι οι ΗΠΑ ξεκίνησαν πρώτες, οπότε ξεκίνησαν πρώτες ε, τη διόρθωση της κατάστασης, πήραν μεγάλες αποφάσεις γρήγορα γιατί είναι μια χώρα, τα ξέρετε αυτά. Ε, και εδώ πέρα στην Ευρώπη είμαστε πίσω. Χρειάζεται ε, ξανά ανακεφαλαιοποίηση πολλών μεγάλων τραπεζών και ελπίζω τα τεστ κοπόσεως που ξεκινάει τώρα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα πραγματικά να λειτουργήσουν. Γιατί, γιατί, ε, τρίτη και τυχερή, τι να πω. Την πρώτη φορά ήταν φεδρή η υπόθεση, δεύτερη, ε, τη δεύτερη φορά εξετάστηκε το δημόσιο χρέος που είχαν στο χαρτοφυλάκιό τους, αυτή τη φορά πρέπει να είναι σοβαρή η διαδικασία, διαφανής και να έχει αξιοπιστία. Όπως ξέρετε εμείς στον ΩΣΑ πιέζουμε για ένα διαχωρισμό, όχι υποχρεωτικό ή τύπου Glass-Steagall, αλλά διαχωρισμό των δραστηριοτήτων Λιανικής ε, Τραπεζικής και Επενδυτικής Τραπεζικής και για ένα ποσοστό μόχλευσης 5% ε, που είναι ψηλότερο από τους κανόνες ε, της Βασιλείας 3. Και τέλος, μέρος απώλειας της εμπιστοσύνης που ανέφερα σχετίζεται με το ότι ο πολίτης βλέπει πως οι πλούσιοι παίρνουν τα λεφτά τους σε φορολογικούς παραδείσους και οι πολυεθνικές δεν πληρώνουν φόρους. Άρα οι μεσαίες τάξεις, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ε, οι εταιρείες που δεν έχουν διεθνείς δραστηριότητες πληρώνουν το λογαριασμό των φόρων κυριολεκτικά. Οι G8 και η G20 έδωσαν έντολη στον ΩΣΑ να εργαστεί ώστε να πάμε σε αυτόματη ανταλλαγή φορολογικών πληροφοριών. Ήδη σήμερα 120 χώρες θα ανταλλάσσουν πληροφορίες κατόπιν αιτήματος. Τώρα πάμε σε ένα πιο φιλόδοξο καθεστώς, πιο αποτελεσματικό, της αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών. 60 χώρες ήδη έχουν δεσμευτεί, μόλις τελείωσε η συνεδρίαση στην ε, Τζακάρτα, 60-62 χώρες και άλλες 50-60 τους επόμενους μήνες, οπότε θα πάμε σε αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών μέχρι το τέλος του επόμενου έτους. Αλλά το πιο σημαντικό, το πιο δύσκολο ζήτημα, η αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών σημαίνει πώς επιβάλλουμε τους, χώρου, τους νόμους κάθε χώρας. Τους δικούς σας νόμους δηλαδή, εδώ πέρα. Το ε, BEPS όμως, δηλαδή η μείωση της ε, φορολογητέας ύλης, Σημαίνει γιατί από την κοινωνία των εθνών ήδη προσπαθούμε να αποφύγουμε τη διπλή φορολογία. Τα καταφέραμε, αλλά δημιουργήσαμε τη διπλή μη φορολογία. Δηλαδή οι πολυεθνικές δεν πληρώνουν πουθενά φόρους. Και τώρα, για πρώτη φορά, κάθε μέλος των G20, είτε είναι η Κίνα, το Μεξικό, η το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γερμανία, όλες οι χώρες έχουν ένα κοινό στόχο. Ότι θέλουν, θέλουν τα λεφτά. Και τώρα μας δόθηκε εντολή να προσπαθήσουμε να αλλάξουμε ουσιαστικά τους κανόνες της διεθνούς φορολογίας. Στην ε, τελευταία συνεδρίαση των G20 στην Αγία Πετρούπολη, ο πρόεδρος Πούτιν είπε πως το θέμα αυτό είναι πιθανώς ότι πιο επαναστατικό έχει γίνει στη διεθνή φορολογία τα τελευταία 100 χρόνια. Αυτό λοιπόν έχετε κατά νου και είναι ένα από τα μεγάλα εκκρεμή ζητήματα. Θα σταματήσω λοιπόν εδώ πέρα και θα δεχτώ σχόλια, ερωτήσεις, ε, ύβρις, ό,τι θέλετε. Ε, βλέπω ότι επιδείξατε διάφορες σελίδες από τις ε, σημειώσεις σας, ε, αλλά με τις ερωτήσεις μας θα σας βοηθήσουμε να χρησιμοποιήσετε αυτές τις σημειώσεις. Ε, βεβαίως στην Επιτροπή, Επιτροπή μας στη ιδιαίτερα για φορολογικά ζητήματα, αλλά όπως σωστά είπατε, διαπιστώθηκε ότι όχι μόνο λείπουν ε, τα έσοδα από τους φόρους σε άλλες χώρες, αλλά και στην Ευρωπαϊκή Ένωση το ίδιο. Και Νομίζω ότι αυτό είναι χρήσιμο για να ασκήσουμε πίεση στις κυβερνήσεις ώστε να αναλάβουν δράση σε τομείς όπου οι ευρωβουλευτέ έχουν ήδη ασκήσει πίεση όχι μόνο κατά τη διάρκεια της τρέχουσας θητεία, αλλά και της προηγούμενε. αλλά εξάλλου και στη δική μου έκθεση για την φοροαποφυγή, φοροδιαφυγή ε, το ίδιο έκανε ο Παύλο Σάλβα, αντιπρόεδρος τη Επιτροπής. Θα ήθελα, Πρόεδρε, να μιλήσω τη γλώσσα μου. Συμφωνώ απολύτως με αυτό που μας είπατε. Θα ήθελα όμως να επανέλθω σε ένα θέμα, αυτό της πίστης. Μας λέτε ότι η στις χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν μηδενική ανάπτυξη κατά μέσο όρο και στην Ισπανία ήταν μείον 4%, μείον 20% ε, ε, σε σχέση με τα προηγούμενα έτη και μείον 50% σε σχέση με την αρχή της κρίσης. Ε, βρισκόμαστε λοιπόν σε αυτή την κατάσταση και θα έπρεπε για να εξέλθουμε από αυτή την κρίση να απελευθερωθεί η πίστη ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ε, η χορήγηση δανείων ε, δηλαδή. Τι μπορούμε να κάνουμε λοιπόν για να αρχίσει να ρέει το χρήμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να υπάρξει ρευστότητα και να απελευθερωθεί ο τομέας της πίστης. Τι μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να πιμπλακεί η κατάσταση σε σχέση τώρα με την ε, συμφωνία που τώρα διαπραγματευόμαστε με τις ΕΙΠΑ για τις επενδύσεις, την TTIP, ε, οι συνάδελφοι αναφέρουν ότι δεν θα πρέπει να συγχέουμε την ε, κατασκοπία με τις εμπορικές ανταλλαγές. Εμπορικέ συναλλαγέ. συγγνώμη. Δεν με... Πιστεύετε λοιπόν ότι θα έχει μεγάλο ειδικό βάρος αυτή η συμφωνία. Πώ ε, τη βλέπετε ακριβώς. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ ε, για την ε, ερώτησή σας. Οι πιστοτικές ροές θα ανακάμψουν όταν επέλθει και η ανακεφαλοποίηση των τραπεζών. Αλλά θα δούμε και περισσότερες πιστοτικές ροές όταν τελικά ολοκληρωθεί η όλη διαδικασία της Τραπεζικής Ένωσης και όταν αποφασίσουμε τελικά ποιος θα επιβλέπει τις τράπεζες, ποιος θα είναι υπεύθυνο ε, για, τη ρύθμιση των τραπεζών και για το πώς θα καταφέρουμε να αντιμετωπίσουμε τις ε, τράπεζες εκείνες που χρεοκοπούν. Πέρα όμως από τα ζητήματα αυτά που είναι ακόμα εκκρεμή, πρέπει να δούμε και το ακόλουθο. Αν θεωρήσουμε ότι μια τράπεζα δεν θα χρεοκοπήσει επειδή θα ανακεφαλοποιηθεί, τότε θα πρέπει να αποφασίσουμε και ποιο θα είναι υπεύθυνο για την ανακεφαλοποίηση αυτή ακόμα και σε προσωρινό επίπεδο. Θα είναι οι κυβερνήσει ή θα υπάρχει ένα κεντρικό μηχανισμό υπεύθυνο για την ανακεφαλοποίηση των τραπεζών. Οι αποφάσει αυτέ είναι σημαντικότατε και πρέπει να ληφθούν το συντομότερο δυνατό προκειμένου να δούμε νέε πιστοτικέ ροέ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό δεν έχει συμβεί ακόμα και όντω υπάρχουν κάποιε τράπεζε οι οποίε κινδυνεύουν και το πρόβλημα βέβαια είναι ότι δεν έχουμε ολοκληρώσει ακόμα τη διαδικασία της ανακεφαλοποίησής τους. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει πάρει κάποιες αποφάσεις προκειμένου να αυξηθεί η ροή των κεφαλαίων, αλλά η πρωτοβουλία αυτή πρέπει να προωθηθεί ακόμα περισσότερο. Του των λεχθέντων, το σημαντικότερο είναι να έχουμε μια γενικότερη σφαιρική τραπεζική ευτεκτονική στην Ευρωπαϊκή Ένωση, προκειμένου να ξέρουν οι τράπεζε ακριβώ τι μπορούν να κάνουν και προκειμένου να αρχίσουν τελικά να δανειοδοτούν. Όσον αφορά τώρα την εμπορική συμφωνία με τι ΗΠΑ. Υπάρχει ένα πρόβλημα εμπορικής φύσης και στη συνέχεια καλούμε να αντιμετωπίσουμε και άλλα προβλήματα όπως η ανεργία, η αυξανόμενη ανεργία, οι αυξανόμενες ανισότητες, το ότι έχουμε πολύ, ασθενή, πολλές πολύ, θεσμικά όργανα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι η κατάσταση είναι γενικότερα αρνητική σήμερα και αποτελεί μια γενικότερη απειλή για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στη συνέχεια έχουμε βέβαια κάποιες τάσεις προστατευτισμού όσον αφορά το εμπόριο, ασθενείς επενδύσεις, συναλλαγματικές ισοτιμίες οι οποίες δεν βοηθούν πάρα πολύ την κατάσταση. Τι βλέπουμε λοιπόν. Αυτό το οποίο πρέπει να κάνουμε είναι να συνεχίσουμε να καταπολεμούμε όλες τις τάσεις εμπορικού προστατευτισμού που αναδύονται αυτή τη στιγμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο προστατευτισμός αυτός σε καμία περίπτωση δεν βοηθά την οικονομική ανάπτυξη, ακριβώς το αντίθετο κάνει. Αν λοιπόν σημειώσουμε επιτυχία στους στόχους μας, αν καταφέρουμε τελικά να προωθήσουμε περισσότερο τις διαπραγματεύσεις και αν καταφέρουμε να έχουμε μεγαλύτερη ολοκλήρωση σε περιφερειακό επίπεδο, θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι από το 50% του παγκοσμίου ΕΠ ένα 30% προέρχεται από το εμπόριο και το υπόλοιπο από τις διεθνείς επενδύσεις και η σημαντικότερη παγκόσμια εταίροι στο εμπόριο και σε επενδύσει είναι οι Ηνωμένε Πολιτείε και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι μια εμπορική συμφωνία ανάμεσα σε αυτέ τι δύο περιοχέ του κόσμου θα καταφέρει να τονώσει πάρα πολύ σημαντικά την παγκόσμια ανάπτυξη. Έχετε έπειτα στη συνέχεια περιφερειακές ολοκληρώσεις εμπορικές σε περιοχές όπως ο Ειρηνικό, με χώρες όπως το Μεξικό, η Κωνσταντίνα κτλ και οι διαπραγματεύσει αυτέ είναι πάρα πολύ σημαντικέ, ιδίω βέβαια για τα κράτη-μέλη του ΩΣΑ. Εμεί είμαστε λοιπόν προφανώ υπέρ τη ε, εμπορική αυτή συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και Ηνωμένων Πολιτειών και θεωρούμε ότι αυτό θα βοηθήσει τόσο την Ευρώπη όσο και του Αμερικάνου σε καθημερινό επίπεδο. Ε, Μια ερώτηση ακόμα κύριε Γενική Γραμματέα. η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων μπορούν να κάνουν περισσότερα πράγματα προκειμένου να έχουμε μεγαλύτερη δανειοδότηση κυρίως προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Είπατε ξεκάθαρα εσεί τι έχει συμβεί μέχρι σήμερα. Τι παραπάνω μπορεί να γίνει όμως στο μέλλον. Αυτή είναι η ερώτησή μου. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα επιτελεί το έργο της αυτή τη στιγμή. Δανείζει χρήματα προς τις ε, μικρομισές επιχειρήσεις, όχι άμεσα όμως αυτές. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων το κάνει αυτό μέσω τραπεζών, μέσω επιμέρους τραπεζών. Το πρόβλημα με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είναι ότι δεν είναι μια κλασική εθνική κεντρική τράπεζα. Παρτίζεται από 18 χώρες και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα λοιπόν στο παρελθόν έχει εργαστεί πάρα πολύ καλά όταν δεν υπήρχε μεγάλη ρευστότητα στο τραπεζικό σύστημα. Δεν έχει όμως την απαραίτητη αρμοδιότητα αυτή τη στιγμή προκειμένου να δώσει μια νέα όθηση στις πιστοτικές αυτές ροές. Την εξουσία αυτή την έχουν τα εθνικά θεσμικά όργανα. και ξέρετε ότι θα πρέπει να συγκλίνουν οι απαραίτητες αντικειμενικές προϋποθέσεις προκειμένου να μπορούμε να έχουμε μια σημαντικότερη δανειοδότηση προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Οι αποφάσει λοιπόν αυτέ εξαρτώνται από τι εθνικέ κυβερνήσει πάρα πολλέ φορέ. Προκειμένου να καταφέρουν να δανειοδοτηθούν περισσότερο οι μικρομεσαίε επιχειρήσει, θα πρέπει να ληφθεί υψηλότερο κίνδυνο και από τι επιχειρήσει αυτέ καθ' αυτέ και από τι εθνικέ τράπεζε που τι χρηματοδοτούν. Ευχαριστώ. Η Ελίζα Φερέιρα από του Σοσιαλιστέ. Ευχαριστώ. Θα μιλήσω πορτογαλικά. Ευχαριστώ το Γενικό Γραμματέα του ΟΣΑ. Θα ήθελα να σας κάνω τρεις ερωτήσεις. Πρώτον, για την Ευρωζώνη. Αντίθετα με τη ΣΥΠΑ, ε, δεν έχει ξεκινήσει η ανάκαμψη στην Ευρωζώνη. Παλεύουμε με ένα ε, ενίο νόμισμα είναι μια μοναδική παγκόσμια εμπειρία αυτό το ενίο νόμισμα. Έχετε προτάσεις, ε, εισηγήσεις ε, σε σχέση με την βέλτιστη λειτουργία αυτής της Ευρωζώνης μετά την κρίση και παραπέμπω σε αυτά που μας είπατε ήδη για την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ασχολείται με τον έλεγχο του πληθωρισμού πέραν αυτού, ποια, ποιο δημοσιονομικό ρόλο μπορεί να παίξει, ποια διδάγματα μπορούμε να αντλήσουμε από την κρίση ε, και πώς μπορεί να μας βοηθήσει ο ΩΣΑ. Δεύτερη ερώτηση, ε, φορολογική παράδειση. Εγώ πιστεύω πως είναι ένα από τα βασικότερα ζητήματα ε, όπου βλέπουμε τη χρησιμότητα του έργου του ΩΣΑ. Εάν ε, δεν ε, καταργήσουμε την φοροαποφυγή και φοροδιαφυγή θα χάσουν οι κυβερνήσεις εντελώς την νομιμοποίησή τους στα μάτια των πολιτών μετά τις περικοπές των μισθών, των συντάξεων. Δεν είναι αφόρητη η κατάσταση τι μπορούμε να κάνουμε για να σταματήσει αυτή η πάγια φοροδιαφυγή των μεγάλων. Ε, μία τρίτη πιο γενική ερώτηση. Ε, ζούμε την εποχή της παγκοσμιοποίησης ε, και είμαστε, είναι μεγάλη αλληλεξάρτηση όλων μας, ε, κυρίως σε περιόδους κρίσης. Λοιπόν, σε παγκόσμιο επίπεδο μπορούμε να συνεχίσουμε με τους θεσμούς που έχουμε κληρονομήσει από τη Συμφωνία Bretton Woods. Μήπως ήρθε η ώρα να αναθεωρήσουμε λίγο τους θεσμούς, τα θεσμικά όργανα που χρησιμοποιούμε σε αυτή την εποχή παγκοσμιοποίησης ώστε να είμαστε πιο οργανωμένοι και να είναι πιο εναρμονισμένη οργάνωση. Ευχαριστώ που με ακούσατε και στα πορτογαλικά. Ευχαριστώ. Ε, το θέμα της Ευρωζώνης, απαντά ο κύριος Σχούρια, ε, στα πορτογαλικά, ε, σχετίζεται με διαρθρωτικά προβλήματα. Ήδη έχουμε εξαντλήσει τις δυνατότητες που έχουμε ως προς την νομισματική πολιτική. Έχουμε φτάσει στα επιτόκια σχεδόν στο 0%. Έχουμε μια δημοσιονομική ικανότητα η οποία έχει σχεδόν εξαντληθεί ως αποτέλεσμα των προσπαθειών που έχουν καταβληθεί για να εξέλθουμε από την ύφεση. Αυτή τη στιγμή προσπαθούμε να μειώσουμε ε, το χρέος και το έλλειμμα. Δηλαδή ε, δεν έχουμε μεγάλη δυνατότητα δημοσιονομικής επέκτασης. Ποιο είναι το ζητούμενο λοιπόν. Είναι να γίνουν διαρθρωτικές αλλαγές, υπάρχουν τα κοινωνικά ζητήματα, τα ζητήματα της πράσινης ανάπτυξης, τα θεσμικά ζητήματα όπως σας έλεγα προηγουμένως. Όταν μιλάω για τα διαρθρωτικά ζητήματα ποια είναι. Μιλάω για την παιδεία, την καινοτομία, τις δεξιότητες. Χρειαζόμαστε περισσότερες δεξιότητες. Χρειαζόμαστε καλύτερη απορρίθμιση επίσης. Σας μίλησα και για τα φορολογικά ζητήματα και την αναθεώρησή τους. Έχουμε περισσότερη φορολόγηση της εργασίας, του κεφαλαίου Αλλά χρειαζόμαστε λιγότερη φορολόγηση της εργασίας. Δεν μπορούμε έτσι να αντισταθμίζουμε την μείωση της φορολόγησης, της κατανάλωσης και της ιδιοκτησίας φόροι που είναι λιγότερο διαρθρωμένοι, αν θέλετε, σε σχέση με τους φόρους ε, στην αγορά εργασίας. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε με την αύξηση των φόρων. Στις περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης διαπιστώνουμε ότι έχουμε την ε, υψηλότερη δυνατή φορολόγηση της εργασίας. Ε, ενώ έχουμε και τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας. Δεν ε, συμβαδίζουν αυτά τα δύο. Δεν μπορούμε να φορολογούμε την εργασία και να θέλουμε να αυξήσουμε την απασχόληση. Δεν γίνεται. Χρειαζόμαστε αναθεώρηση του ρόλου της ΕΚΤ. Ε, η ΦΕΔ δεν έχει τόσο μεγάλο περιθώριο ελιγμών που αγοράζει δημόσιο χρέος, όπως και στην Ιαπωνία εξάλλου με ε, τις 18 ε, χώρες ε, στην Ευρωζώνη μπορεί να βοηθήσει η έκτη να σταθεροποιηθεί η κατάσταση όχι μόνο μέσα από τα επιτόκια γιατί ξαναλέω δεν, μπορεί, δεν περιορίζεται μόνο στην εξαγορά ε, χρέους. Για το θέμα της ε, φοροαποφυγής, φοροδιαφυγής και φορολογικής απάτης θα πρέπει να αναχαιτιστεί πάση θυσία. Αυτό σχετίζεται με την παγκόσμια αρχιτεκτονική. Πιστεύω πως ε, η ομάδα G20 η G, μάλλον η ομάδα G8 δεν επαρκεί η ομάδα G20 είναι αυτή που πλησιάζει περισσότερο μια λειτουργική αρχιτεκτονική σε παγκόσμιο επίπεδο σε σχέση με ε, τους παραδοσιακούς θεσμούς, αυτούς που κληρονομήσαμε τον Bretton Woods. Ακόμη και ο ΩΣΑ πρέπει να μετεξελιχθεί, πρέπει να τροποποιηθεί, να προσαρμοστεί ε, στα νέα δεδομένα ε, άσχετα με το τι θα κάνουν οι μεγάλες αναπτυσσόμενες χώρες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρόεδρος, ευχαριστώ που ε, σας ζήτησα να συντομεύσετε, γιατί αν ξεφύγουμε από τη χρονοθυρίδα την πεντάλεπτη θα απογοητευτούν τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής. Ε, ήρθε η σειρά των φιλελευθέρων εγώ πρέπει να μιλήσω γιατί δεν υπάρχει κανένας άλλος. Ε, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τη δουλειά που έχει κάνει ο ΣΑΜ για τη διάβρωση της φορολογικής βάσης ε, και την ε, μεταφορά ε, και πλημελή εκτίμηση των στοιχείων ενεργητικών των θηγατρικών εταιριών των μεγάλων ομίλων. Είδαμε ότι μπορούμε να επιδιώξουμε καλύτερη δημοσιοποίηση των πληροφοριών κατά της επιθετικής φορολογικής πολιτικής των μεγάλων ομίλων και χωρίς να ντρέπομαι καθόλου αντέγραψα τα πορίσματα της δικής σας δουλειάς και τα έβαλα στην έκθεσή μου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. η πλειοψηφία της Επιτροπής ε, έχει ε, πάρει τη δική μου θέση και ε, δεν μπορώ να πω το ίδιο για την Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων. Τέλος πάντων, δεν πρέπει να τρεπόμαστε που σας ακολουθούμε. Κάποιος πρέπει να έχει τον ηγετικό ρόλο για τα φορολογικά ζητήματα και σας άκουσα με προσοχή. για το θέμα της διαφάνειας επανέρχεται συνέχεια αυτό το ζήτημα των εταιριών που καταγγέλουν την ε, έλλειψη δημόσιας διαφάνειας ε, κατά τη διαστολή με την επιδίωξη της διαφάνειας μόνο σε φορολογικά ζητήματα μέσω δημοσιοποίησης πληροφοριών από πλευράς τους. Οπότε... Ε, μας κατηγορούν ότι αυτό που επιδιώκουμε είναι να, αναδειχθούν, να αναδειχθεί η έλλειψη δημοσιοποίησης σε ποινικό αδίκημα μόνο και μόνο για να μπορεί να διωχθεί από κάποια δημόσια αρχεία. Εσείς τι λέτε. Ε, πιστεύετε ότι υπάρχουν, ε, ε, υπάρχει, έχουν δίκιο, δηλαδή καλά κάνουν και προσπαθούν να μας εμποδίσουν. Ευχαριστώ. Απάντηση. Κοιτάξτε, το μπέψτε το, το σχέδιο δράσης μας για την διάβρωση της φορολογικής βάσης είναι ένα από τα μεγαλύτερα και πιο ρηξικέλευτα εγχειρήματα που έχουμε να λάβει στον ΟΣΑ. Κάποιοι μας λένε ότι ναι, συνιστά ρήξη σε σχέση με το παρελθόν και άρα καλά κάνετε και είσαστε τόσο φιλόδοξοι. Ε, κοιτάξτε, ε, με τους φορολογικούς παραδείσους ε, τι μπορούμε να κάνουμε, ότι ε, να μην μπορούν να κρυφτούν πουθενά. Αυτό μπορούμε να το επιδιώκουμε μόνο για τους ιδιώτες. Και τι κάνουμε, επιβάλλουμε το νόμο και λέμε πρέπει να πληρώνετε τους φόρους σας εδώ. Όμως, Ξέρετε τι έχουμε κάνει, το, έχουμε θεσπίσει φορολογικούς κανόνες βάσει των οποίων είναι νόμιμο, είναι νόμιμο να μην πληρώνει μια εταιρεία τους φόρους, καταλαβαίνετε. Πρέπει να τροποποιήσουμε λοιπόν την ε, νομοθεσία σε όλες τις χώρες που εμπλέκονται σε αυτό το εγχείρημα με τρόπο ώστε να υπάρξει μια ομοιογενής ομοιόμορφη προσέγγιση. Βεβαίω, δεν μπαίνουμε στα χωράφια των κρατών. Ε, ε, η διεθνική κυριαρχία ισχύει και παραμένει στα φορολογικά ζητήματα. Γι' αυτό έχουμε στραφεί προ την δημοσιοποίηση πληροφοριών και πάλι να μην επιτρέψουμε να μην έχουν πουθενά να κρυφτούν. Και πάλι ε, οι εταιρείε σας λέω, εάν ε, μία εταιρεία παράγει στην επικράτεια ενός κράτους ε, και δημιουργεί πλούτο και αποκομίζει κέρδη και δημιουργεί θέσεις απασχόλησης στην επικράτειά σας, πάρα πολύ ωραία. Για τον πλούτο όμως που παράγει πρέπει να πληρώνει και τους φόρους. Θα ήθελα επίσης να απαντήσω στο πολύ συγκεκριμένο σας ερώτημα. Αυτή τη στιγμή στην ε, Φορολογική Επιτροπή του ΟΣΑ αλλά και της ομάδας G20 ε, η Ινδία, η Βραζιλία, η Κίνα, όλοι συμμετέχουν σε αυτήν την ομάδα εργασία. Δεν έχουμε αποκλείσει κανέναν. Λοιπόν, και θα καταλήξουμε σε μία σειρά προτάσεων ε, περίπου σε 18 μήνες. Σας ενθαρρύνω αν ναι, και άμα μου επιτρέπετε να τους πω να έρθουν εδώ να σας τα πούνε και οι ίδιοι. Όταν βλέπετε κάποια συγκεκριμένη φρασιολογία, κάποια συγκεκρι... κάτι που θέλετε να εισαχθεί σε αυτή την νομοθεσία πρέπει να μας το πείτε. Ένα όμως θα είναι το πρότυπο, δεν μπορούμε να έχουμε 150 γιατί θα πάνε θα κρυφτούν στο πλέον ευνοϊκό και χαμηλότερο για αυτούς πρότυπο εάν δεν το κάνουμε αυτό. Οπότε... μόνο αν έχουμε ένα κοινό μέτωπο και ένα κοινό ε, πρότυπο θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Χρειαζόμαστε τη δική σας την υποστήριξη για να τα καταφέρουμε. Διαφάνεια, δημοσιοποίηση πληροφοριών, ναι και σε κάποιες χώρες ε, τι λένε, χρησιμοποιούν αυτό το κακό πρόσχημα, μας λένε όχι δεν ε, είναι καλή η δημοσιοποίηση, ε, δεν είναι καλή η διαφάνεια, δεν είναι πολύ κακή άμυνα. Η δημοσιοποίηση και η διαφάνεια πρέπει να είναι ο κανόνας, πρέπει να είναι το εφαρμοστέο πρότυπο και μόνο έτσι ε, θα αντιμετωπίσουμε ε, τον επιθετικό φορολογικό σχεδιασμό και την ε, πλημελή εκτίμηση των στοιχείων ενεργητικού των εταιριών στα πλαίσια των ομίλων. Για το transfer pricing τώρα, αυτό το ζήτημα ξέρετε τι συμβαίνει. Εάν δεν υπάρχει μέτρο σύγκρισης, πώς μπορούμε να αποφασίσουμε τίποτα, κάτι σκεφτείτε πόσα μαγαζιά Apple έχετε, πόσα μαγαζιά Starbucks, ε, πόσα πόσες θυγατρικές ε, ε, υπάρχουν σε αυτές τις μητρικές, σε πόσες, ε, σε πόσες χώρες δραστηριοποιούνται. Δημιουργείται δηλαδή μια νέα κατάσταση όπου κυρίως στον τομέα της πληροφορικής επιτρέπεται παρουσία, πανταχού παρουσία κάποιων εταιριών και πώς εμείς θα προσαρμόσουμε την νομοθεσία για να το αντιμετωπίσουμε αυτό. Γι' αυτό σας λέω ότι χρειαζόμαστε τη δική σας βοήθεια. Ας ενώσουμε τις προσπάθειες Πρόεδρος, ε, ευχαριστώ. Ο στόχος είναι να σκάψουμε για να βρούμε τις πληροφορίες ε, πρώτα για να μπορέσουμε να πράξουμε και στη συνέχεια. Αλλά αυτή περίφημη αρχή arm's length ε, ε, κολλάει στο ότι κάποιοι έχουν πολύ μακρύτερο χέρι από τους άλλους. Ε, ο Ντέρκ από τους συντηρητικούς. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε και τον κύριο Γκουρί επίσης να ευχαριστήσω για τα αισιόδοξα στοιχεία τα οποία μας έδωσε. Στις οικονομικές προβλέψεις που δημοσίευσε ο ΣΑ κάνει κάποιες προτάσεις. Λέει ότι οι Ηνωμένε Πολιτείε θα πρέπει να συνεχίσουν με την επεκτατική νομισματική πολιτική τους και ότι θα πρέπει να τερματιστούν κάποια στοιχεία της νομισματικής αυτής πολιτικής. Από την άλλη όμως λέτε ότι θα πρέπει να επεκταθεί περισσότερο η νομισματική αυτή πολιτική αν οι αποπληθωριστικές πιέσεις γίνουν όλο και μεγαλύτερες. Λέτε λοιπόν ότι η ΦΕΤ θα πρέπει να τυπώσει λιγότερα δολάρια, ενώ η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα πρέπει να τυπώσει περισσότερα ευρώ. Εσείς κύριε Γκουρία γνωρίζετε πώς εξελίχθηκαν τα πράγματα στα πλαίσια του Επαναστατικού Κόμματος του Μεξικού, στο οποίο συμμετείχατε και το θεωρώ ότι είναι το αντίστοιχο του δικού μας Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή διανύει μια πολύ δύσκολη κατάσταση και βλέπουμε ότι ιδίω εξαιτία κάποιων φαινομένων όπως η ανεργία μπορούμε να έχουμε πολύ δυσμενείς επιπτώσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν να γνωρίζουμε αν η πολιτική την οποία εσείς προτείνετε θα έχει τελικά κάποιες αρνητικές επιπτώσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αν οι δικές σας προτάσεις, οι δικές προτάσεις όσον αφορά την νομισματική πολιτική μπορούν τελικά να βοηθήσουν την Ευρωζώνη και αν τελικά θα οδηγήσουν σε μεγαλύτερη οικονομική ανάπτυξη και σε πάταξη της ε, ανεργίας. Ο λόγος, σας ευχαριστώ για την ερώτησή σας, ο λόγος για τον οποίο έχουμε διαφοροποιημένη προσέγγιση στις νομισματικές πολιτικές είναι γιατί οι ίδιες οι οικονομικές υπεριφέρειες βρίσκονται σε διαφορετική χρονική στιγμή, σε διαφορετική περίοδο. Οι Ηνωμένε Πολιτείες ξεκίνησαν μια πάρα πολύ επιθετική κίνηση με χαμηλά επιτόκια και στη συνέχεια άρχισαν να χαλαρώνουν την νομισματική τους πολιτική από ποσοτικής πλευράς και βρίσκονται πλέον στο τρίτο σχετικό στάδιο. Η κεντρική τους τράπεζα αγοράζει το χρέος της ίδιας της χώρας προκειμένου να καταφέρει να μειώσει τα επιτόκια τόσο βραχυπρόθεσμα αλλά και μακροπρόθεσμα κάνει τις απαραίτητες διεργασίες όπου αγοράζει μακροπρόθεσμα στοιχεία του ενεργητικού προκειμένου τα επιτόκια να παραμείνουν χαμηλά σε μια, για μια διετή, τριετή περίοδο. Αυτό είναι θετικό γιατί βλέπουμε ότι υπάρχουν και άλλες κεντρικές τράπεζες που ακολουθούν το παράδειγμα αυτό όπως η Κεντρική Τράπεζα της Αγγλίας ή της Ιαπωνίας. Ουσιαστικά κατά αυτόν τον τρόπο οι τράπεζες αυτές, οι κυβερνήσεις αυτές κατάφεραν να μειώσουν τη σοβαρότητα της κρίσης, κατάφεραν να κρατήσουν τα επιτόκια τεχνητά πολλές φορές, πολύ χαμηλά, προκειμένου να καταφέρουν να κάμψουν γρηγορότερα από την οικονομική κρίση. Η ΦΕΤ πάντως δεν μπορεί να, να συνεχίζει να βάζει στον κρατικό ισολογισμό ένα τρισεκατομμύριο δολάρια σε τήσια βάση και ξέρετε ότι χρειάστηκε να αντιμετωπίσουν μια εξαιρετική κατάσταση στην αρχή και αυτή τη στιγμή λένε ότι θα αρχίσουν να μειώνουν τις αγορές στοιχείων του ενεργητικού. Ουσιαστικά οι αγορές τους αυτές στο μέλλον, αντί να είναι 85 εκατομμύρια το μήνα, θα γίνουν 75, 70, 60 και το καθεξής. Ουσιαστικά αυτά είναι θετικά νέα. Λένε σιγά σιγά ότι αρχίσουν και μειώνουν το φάρμακο, αρχίζουν και μειώνουν την κορτιζόνη αν θέλετε. Αυτό σημαίνει ότι η κατάσταση αρχίζει σιγά σιγά να, ομαλοποιεί, να εξομαλύνεται. Ο ασθενής όμως ενδεχομένω να ζητήσει περισσότερο φάρμακο γιατί πολύ φοβάται ότι τελικά μπορεί να εκτεναχθούν πάλι τα επιτόκια, ότι μπορεί να μην εξελιχθεί πάρα πολύ θετικά η κατάσταση. Η σταδιακή αυτή μείωση που βλέπουμε από πλευρά κεντρική τράπεζα τη Αμερική ήταν προβλέψιμη, αναπόφευκτη και θα έλεγα ότι ήταν και ευκταία, διότι καταδεικνύει τελικά ότι μπαίνουμε σιγά σιγά σε μια ομαλή κατάσταση. Και η ομαλή αυτή κατάσταση θα πρέπει να είναι ο κανόνα, αν θέλετε. Τώρα, τι γίνεται στην Ευρώπη. Στην Ευρώπη δεν έχουμε φτάσει ακόμα σε αυτό το στάδιο. Γιατί, γιατί η οικονομική ανάπτυξη στην Ευρώπη, όπως σας είπα, είναι πάρα πολύ χαμηλή, είναι ουσιαστικά αρνητική όσον αφορά την Ευρωζώνη ακόμα για φέτος. Θα δούμε μια πολύ ήπια οικονομική ανάκαμψη για το 2014 Συνεπώς χρειαζόμαστε ακόμα χαμηλά επιτόκια στην Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να παγιοποιήσουμε περισσότερο τη διαδικασία της ανάκαμψης. Για 15 χρόνια η Ιαπωνία από την άλλη έχει φλερτάρει με τον αποπληθωρισμό. Στοχεύει στο να δημιουργήσει ένα πληθωρισμό 2% στο μέλλον. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο 0,9% το πολύ. Στην Ιαπωνία λοιπόν έχουν μια πολύ επιθετική νομισματική πολιτική και προσπαθούν να διπλασιάσουν τα χρήματα που ρίχνουν στην αγορά σε δύο έτη. Θα φτάσουν τα 2 τρισεκατομμύρια γεν τα 270 τρισεκατομμύρια γεν τα επόμενα χρόνια. Χρειάζονται τα χρήματα αυτά. Πρέπει να καταφέρουν να τονώσουν την οικονομία τους. Γι' αυτό κάνουν και από δημοσιονομικής και διαρθρωτικής πλευράς. Βλέπετε πάντως στις διαφορετικές αυτές γεωγραφικές περιοχές, τα διαφορετικά στάδια στα οποία βρισκόμαστε. Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο εμεί συστήνουμε διαφορετικές νομισματικές πολιτικές με βάση τη γεωγραφική ζώνη, με βάση τις οικονομικές ανάγκες που υπάρχουν στις περιοχές αυτές και με βάση την εξέλιξη της οικονομίας αυτών των περιοχών. Σας ευχαριστώ για τους πράσινους ο Σβεν Γίγκολτ. Καλημέρα. Κύριε Γκουρία. Ωραία είναι να ακούμε κάποια πράγματα που είπατε για την ρύθμιση των χρηματαγορών. Α! Και για γερμανικά καταλαβαίνετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτά τα οποία είπατε τελευταία και δημοσιεύσατε για την κατάσταση του τραπεζικού συστόματος για την Ευρώπη και για αυτό το οποίο είπατε για τις τράπεζες, για την ανάγκη ισχυρότερου διαχωρισμού, εγώ έχω μια άλλη ερώτηση όσα. Ήμουν πολύ μικρός όταν ε, πρώτο άκουσα, για συνάντησα τον Τζέφρι Owens. ήταν τότε διατεθειμένος να μιλήσει με ΜΚΟ για το θέμα της ε, φορολογικής πολιτικής και φορολογικής συνεργασίας και μας προξένηξε έκπληξη το ότι ο συνεργα... η συνεργάτης του, η Καρολάιν Σίλμπερστάιν, έφυγε από τον ΩΣΑ για μια δουλειά σε δικηγορικό γραφείο ονόματι Baker McKinsey που έδινε συμβουλές ε, στην Amazon για το transfer pricing και μετά η Mary Bennett επίσης ε, πήγε στην ίδια εταιρεία απευθείας από τον ΩΣΑ και μετά από 20 χρόνια ο ίδιος ο Jeffrey Owens πήγε στην Ernst Young η οποία διαφημίζει ανοιχτά, σας το διαβάζω. Η προηγούμενη θέση του Τζέφρι ως ε, διευθυντού του Κέντρου Φορολογίας και Διοίκησης του ΩΣΑ του έχει δώσει μια μοναδική διεθνή εμπειρία για την φορολογική πολιτική και ζητήματα φορολογικής πολιτικής. Ε, για πάνω από 20 χρόνια ήταν υπεύθυνο ε, για το θέμα αυτό στον ΩΣΑ. Έτσι διαφημίζει ε, η Ernst Young ε, την περίπτωση αυτή. Όταν κάποιος έχει, δημοσιεύσει, έχει συσσωρεύσει αυτή την εμπειρία, ποιο μηχανισμό έχετε για να μην ε, προκύπτει αυτή η σύγκρουση συμφερόντων. Δηλαδή αυτά τα οποία απέκτησε αυτός ο άνθρωπος ως εμπειρία προς το δημόσιο συμφέρον να τα πουλάει σε μια εταιρεία τι ε, διδάγματα αντλείται για να μην αλλάζουν πλευρά αυτοί οι άνθρωποι έτσι, και να μην, υπάρχει, να μην υπάρχουν αυτά τα αντικρώμενα συμφέροντα. Σας ευχαριστώ. Είναι σημαντικό αυτό το ζήτημα, δηλαδή πώς συνδυάζουμε το δικαίωμα των ανθρώπων μετά από δεκαετία ε, δουλειάς ε, σε ένα διεθνή οργανισμό ή στο δημόσιο το δικαίωμά τους να πάνε να εκμεταλλευτούν τις γνώσεις τους στον ιδιωτικό τομέα και ταυτόχρονα να αποφύγουν αυτό το οποίο λέτε την, ε, τα συγκρόμενα συμφέροντα. Έχουμε κάποιους κανόνες, ε, κάποιες υποχρεωτικές περιόδους ε, που πρέπει να παρέλθουν, οι οποίες διορίες έγιναν σεβαστές Και βεβαίως οι περιπτώσεις αυτές ήταν ε, χρήσιμες γιατί μας βοήθησαν να εκπαιδεύσουμε και κάποιους ανθρώπους. Τώρα όμως πρώτα απ' όλα να σας συγχαρώ και δεύτερον να πω πως οι τελευταία οι κανόνες έγιναν πιο αυστηροί εδώ πέρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση για συγκρόμενα συμφέροντα Κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον και νομίζω είναι υποδειγματικοί οι κανόνες. Τους εξετάζουμε προσεκτικά για να δούμε το εάν μπορούμε να τους μιμηθούμε. Είναι μόνιμο αυτό το ζήτημα. Στη ΣΥΠΑ, παραδείγματο χάρη, βλέπετε ότι υπουργού οικονομικών πηγαίνουν σε τράπεζε μετά. Τραπεζίτες γίνονται υπουργοί οικονομικών. Και είναι το πιο φυσιολογικό πράγμα. Έτσι παίρνουμε τον κύριο Ρούμπιν, τον κύριο Πόλσεν από τη Goldman Sachs και μετά γίνονται Υπουργοί Οικονομικών, όπου θα εποπτεύουν τις τράπεζες, έτσι. Και το ζήτημα είναι... Δεν, δεν τίθεται καν. Οι δε υποχρεωτικές περίοδοι που πρέπει να παρέλθουν είναι σύντομες. Αλλού είναι μεγαλύτερες και υπάρχουν περισσότερες προφυλάξεις πρέπει να προσέξουμε το ζήτημα αυτό και πραγματικά εκτιμώ το ότι το αναφέρατε. Στον ΩΣΑ δεν ανησυχούμε μόνο για αυτό το θέμα ε, γιατί βεβαίως ε, πρέπει αυτά που λέμε να τα κάνουμε κιόλας αλλά γιατί συνεργαζόμαστε με κράτη για να καταπολεμήσουμε τις δωροδοκίες σε διεθνείς συναλλαγές για να έχουμε κάποια κάποιες ε, ηθικές ε, διατάξεις ε, όσον αφορά τις δημόσιες προμήθειες, τα ζητήματα εκεί των λεγόμενων Ολλανδικών δημοπρασίων. Δεν ξέρω γιατί όλα αυτά τα κόλπα λέγονται Ολλανδικά. Έχουμε τις κατευθυντήριες γραμμές, έχουμε και τους, τα εθνικά σημεία επαφής που αφορούν και ζητήματα ηθικά αλλά και ανθρωπινών δικαιωμάτων όταν κατέρευσε το κτίριο στο Μπαγκλαντές ε, είχαμε μια συνάντηση στον ΩΣΑ όπου μεταξύ άλλων φέραμε κάποιες εταιρείες ε, και τώρα βελτιώθηκαν τα πράγματα οπότε είναι σημαντικό σημαντικό το το αναφέρατε πράγματι επαγρυπνούμε και μια που είστε πράσινος θα ήθελα να σας ζητήσω να διαβάσετε και την διάλεξή μου στο London School of Economics ε, που λέγεται πηγαίνοντας προς μηδενικές εκπομπές. Σας ευχαριστώ, αλλά θα αυστηροποιήσετε τους κανόνες ή όχι. Θα διαβάσω την ομιλία σας αν μου υποσχεθείτε ότι θα κάνετε πιο αυστηρούς κανόνες. Όπως σας είπα, το εξετάζουμε και, αυτά, και το τι κάνετε εσείς εδώ πέρα και πάντα προσπαθούμε να αυστηροποιήσουμε τους κανόνες, αλλά να είναι και πρακτική και σκληρή και το κυριότερο διαφανής. Γιατί πρέπει να αποφύγουμε βεβαίως τη σύγκρουση συμφερόντων, αλλά και την εντύπωση τέτοιων αντικρώμενων συμφερόντων. Γιατί βεβαίως αυτό βλάπτει και την αξιοπιστία Ενό διεθνού οργανισμού. Η πρόεδρος. Άρα λέτε δηλαδή ναι εάν μπορούμε. Λοιπόν, όχι Σφεν. 7 λεπτά αφιέρωσαμε ήδη λόγω κάποιου λάθους δεν έδωσα τον λόγο στον συντονιστή του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος θα πάρει λοιπόν τώρα τον λόγο ε, προφανώς ε, ως ε, Παριζιάνος ενδιαφέρεται για τον ΩΣΑ Ζαν Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Επιτρέψτε μου να αρχίσω με ένα αστιάκι. Εάν δεν κάνω λάθος, είναι στο κάστρο Ντελαμιέτ η έδρα του Όσα. Οπότε, εντάξει, καλά όλα αυτά, αλλά ας κάνει και κάτι από αυτά που λέει ο Όσα. Ε, μιλούσατε για φορολογικά ζητήματα, αλλά είναι λίγο σχιζοφρενικά όλα αυτά. Άλλα λέμε, άλλα κάνουμε ο της 14 ε, Νοεμβρίου 2013, πριν από λίγες μέρες, ε, δημοσίευσε ε, μία έκθεση που τυκλοφορεί το «Η Γαλλία ε, δίνει μια κίνηση στην ανταγωνιστικότητα. Ε, και ε, μεγάλο μέρος της έκθεσης ήταν αυτά τα ζητήματα. Βεβαίως είναι γενικές οι προτάσεις που κάνατε και επευκαιρία θα ήθελα να σας ρωτήσω τι πιστεύετε για το νομοσχέδιο φορολογικής μεταρρύθμισης που ξάφνιασε τους πάντες ακόμη και τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Τι πιστεύετε ότι αν περάσει στην πράξη θα έχει μια φορολογία που θα μας οδηγήσει σε μεγαλύτερη κοινωνική δικαιοσύνη και μεγαλύτερη ανάπτυξη. απάντηση. Ευχαριστώ. Ήμουν με τον πρόεδρο Ολάντε στις 8 ε, Νοεμβρίου, δηλαδή έξι ημέρες πριν την παρουσίαση του φακέλου που σας δείχνω. Ε, Επανεκκίνηση της ανταγωνιστικότητας. Αυτός είναι ο τίτλος. η πορεία προς μια καλύτερη πολιτική. Και δώσαμε ένα αντίτυπο και στην ε, κυρία Μέρκελ ε, για την Ευρωζώνη. Ήταν και ο Πάσος Κουέλιο εκεί, ήρθε και μας βρήκε εκεί στο Σατόν Λαμιέτ και του δώσαμε τον ίδιο φάκελο γιατί συνήθως ε, τέτοια ε, ε, έγγραφα παράγουμε, τέτοιου φακέλου όπω αυτό που θα δώσουμε για την Ελλάδα αύριο είναι πλήρης ε, είναι, είναι πλήρης ο φάκελο. Ε, και πέρα από αυτέ τι ε, ενδελεχείς μελέτε έχουμε και τι ειδικότερε, όπω αυτή στην οποία αναφέρεστε και έχουμε στατιστικά στοιχεία και συστάσει για 12, 13, 15 ζητήματα κέρια σημασία για το υποεξέταση θέμα. Λοιπόν, για την ανταγωνιστικότητα τι είπαμε στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. μιλήσαμε για την έρευνα και για την καινοτομία, για το ρυθμιστικό πλαίσιο πλαίσιο για ένα αποτελεσματικότερο δημόσιο τομέα, για τη μεταρρύθμιση του φορολογικού συστήματος ε, υπέρ της απασχόλησης και των επενδύσεων, ε, βελτίωση της, ε, των επιδόσεων του εκπαιδευτικού συστήματος, επαγγελματική κατάρτιση. 32 δις δαπανείτε εσείς στην Γαλλία για την επαγγελματική κατάρτιση. Μόνο το 12% πηγαίνουν σε αυτούς που ψάχνουν να βρουν μια δουλειά. Ε, και αυτό το ποσό ισούται με αυτό που δαπανείται για τα επιδόματα ανεργίας. Είναι πελώριο αυτό το ποσό. 32 δις, 32 δις πρέπει να ε, ε, γίνει νέος καταμερισμός αυτών των κονδυλίων. αγορά εργασίας και το θέμα της προσθέμενης αξίας, η θέση της Γαλλίας στην, ως προς την αξία του, του ΑΕΠ και τα λοιπά. Μιλήσαμε με ε, τους εκπροσώπους της ε, Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, ε, της Παγκοσμίας Τράπεζας, με διάφορους τέλος πάντων και τους παρουσιάσαμε αυτή τη μελέτη. Είναι η πέμπτη που δίνω στον κύριο Ολάντ. Έδωσα την πρώτη Του έδωσα την πρώτη στο Λόσα Κάμπος ε, ε, με την επαύριο ε, των εκλογών όταν ανέλαβε το αξίωμά του. Λοιπόν, μου είπε ότι δεν συμφωνώ 100% με την έκθεση, αλλά συμφωνώ σε μεγάλο μέρος και νομίζω ότι θα συμφωνήσουν και οι κοινωνικοί εταίροι, θα δώσουμε την ε, δέουσα συνέχεια σε αυτή την έκθεση. Ε, είμαστε δημοκρατικοί, έτσι συνομιλούμε με τους ε, ηγέτες και όχι μόνο με τη Γαλλία, με το Μεξικό, με διάφορες χώρες. Του δώσα και ένα πιν, μια κονκάρδα. Νομίζω ότι αυτό που χρειαζόμαστε είναι επικοδομητικός διάλογος με τους ηγέτες. Ε, ναι, αλλά πρέπει να φροντίσετε να μην, να μην τη χάσει την έκθεση. Αφού την, ε, την, ε, του έχετε δώσει 4-5 εκθέσεις, καταλαβαίνετε δεν είστε και πολύ αποτελεσματικός, δεν είναι πολύ αποτελεσματική μέθοδος που προκρίνετε. Ε, σας ευχαριστώ, Άννη για τους σοσιαλιστές. Thank you very ε, σε ευχαριστώ, Σάρον. Φαντάζομαι δεν μιλάτε ελληνικά, κύριε Γενική Γραμματέα. Λίγα ελληνικά, μάλιστα. Θα ήθελα να επανέλθω στα όσα είπατε στην εισαγωγή σας, τα οποία μας εμπνέουν πολύ, αλλά δεν είναι πάρα πολύ αισιόδοξα. Αναφερθήκατε σε τέσσερα κληροδοτήματα της οικονομικής κρίσης, Αναφερθήκατε στην χαμηλή ανάπτυξη, στην υψηλή ανεργία, στο ότι υπάρχουν ανισότητες όσον αφορά το εισόδημα και ότι μειώνεται, ότι έχουμε μια πολύ σημαντική απώλεια της εμπιστοσύνης του κοινού προς τις πολιτικές μας. Είναι πολύ σημαντικά τα τέσσερα αυτά στοιχεία και δεν αναφερόμαστε παρκώς αυτά. Επίσης, περιγράψατε μια κατάσταση όπου βλέπουμε ότι είναι πάρα πολύ χειρότεροι σε κάποιες χώρες οι οποίες υπόκεινται σε ένα πρόγραμμα λιτότητας, όπως η Ελλάδα για παράδειγμα. Είναι η έκτη συνεχής χρονιά ύφεσης, πάρα πολύ ψηλή ανεργία στη χώρα μου, πολύ σημαντικές οι ανισότητες όσον αφορά τις αποδοχές, το εισόδημα και πολύ επικίνδυνη η απώλεια της εμπιστοσύνης του κοινού προς την κυβέρνηση, προς τις πολιτικές εφόσον προτείνεται κάποια μέτρα για την αντιμετώπιση της υφιστάμενης κατάστασης, πιστεύω ότι ε, πρέπει να λάβουμε υπόψη μας και το εξής. Κάτι το οποίο έχει να κάνει με την υφιστάμενη κατάσταση και η ερώτησή μου είναι η ακόλουθη. Η καταθλιπτική αυτή κατάσταση την οποία μας περιγράψατε ήταν τελικά αναπόφευκτη. Ήταν ε, μια αναπόφευκτη συνέπεια των ε, αποφάσεων που ελήφθησαν για την αντιμετώπιση της κρίσης ουσιαστικά γίνανε κάποια στρατηγικά λάθη στην συνταγή αυτή την οποία αποφασίσαμε να εφαρμόσουμε και σας θέτω το ερώτημα αυτό γιατί πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε αν τελικά έχουμε μάθει κάτι από τα λάθη μας, αν έχουμε αγγλίσει κάποια διδάγματα από τα σφάλματα αυτά εφόσον έγιναν σφάλματα και θα πρέπει να γνωρίζουμε αν ο συνδυασμός πολιτικής που εφαρμόζουμε αυτή τη στιγμή στην Ευρωζώνη, ιδίω στις ε, χώρες ε, του Μνημονίου, αν όντως ο συνδυασμός αυτός πολιτικής είναι σωστός. Αν τελικά δηλαδή εφαρμόζουμε όντως μέτρα τα οποία θα βοηθήσουν την οικονομική ανάπτυξη, θα μειώσουν την ανεργία, ιδίως την ανεργία των νέων, θα αντιμετωπίσουν τις ανισότητες στο εισόδημα και ουσιαστικά θα βοηθήσουν στην ανάκτηση της εμπιστοσύνης του κοινού, της κοινή γνώμης. Εσείς εκτιμάτε ότι η Ελλάδα θα έχει χαμηλότερη ανάπτυξη από ό,τι ε, προβλέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή οι ελληνικές αρχές. Θα μπορούσατε να μου δώσετε κάποιες ε, περισσότερες πληροφορίες για το πού τελικά έχετε βασίσει, πού βασίζεστε για αυτές τις εκτιμήσεις σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι σας έχει δοθεί το αντίγραφο αυτό, το οποίο το ονομάζουμε ο κροκόδιλος και το λέμε έτσι γιατί το κόστος εργασίας της Ελλάδας, της Γαλλίας, της Ιταλίας της Ιρλανδίας, της Ισπανίας, της Γερμανίας ακολουθούν αυτή την πορεία. Για 15 χρόνια. Για όλες αυτές τις χώρες ισχύει αυτό το πράγμα. Μου λέτε για ποιο λόγο φτάσαμε στην κατάσταση αυτή, για, ποιο λόγο, για λόγο πρέπει να κάνουμε προσαρμογές, για ποιο λόγο είναι τόσο επώδυνη η προσαρμογή. Εδώ και 15 χρόνια έχουμε μισθούς υψηλότερους από την παραγωγικότητα. Στη Γερμανία για 15 χρόνια έχουμε μία παραγωγικότητα υψηλότερη από τους μισθούς. Και βλέπουμε ότι όλα αυτά συμβαίνουν ενώ το νόμισμα παραμένει το ίδιο, όλες οι υπόλοιπες οικονομικές συνισταμένες παραμένουν οι ίδιες και οι επενδύσεις επίσης. Κατά αυτόν τον τρόπο βλέπετε ότι υπάρχει ένα τεράστιο χάσμα και το χάσμα αυτό παρομοιάζεται με το στόμα του κροκόδιλου. Τι συμβαίνει λοιπόν αυτή τη στιγμή. Στην Ισπανία έχουμε ένα 10% έλλειμμα στην Ισπανία. Έχετε εδώ πέρα σελίδα 25 όλα αυτά τα δεδομένα. Στην Πορτογαλία επίσης έχουμε 10% έλλειμμα. Στην Ιταλία επίσης, στην Ισπανία 10%. Πού βρίσκονται όλες αυτές οι χώρες αυτή τη στιγμή. Όλες αυτές οι χώρες έχουν μηδενική ανάπτυξη όσον αφορά τους τρέχοντες λογαριασμούς. Ξέρετε ότι έχει γίνει μια τεράστια προσαρμογή όσον αφορά το κόστος εργασίας. Και αυτό γιατί αρχίζει σιγά σιγά ο κροκόδιλος να κλείνει τελικά το στόμα του. Αρχίζουν οι τάσεις αυτές που είχαμε δει στο παρελθόν να προσαρμόζονται σιγά σιγά και η Γερμανία και αυτή σιγά σιγά αρχίζει να αυξάνει τους μισθούς της και ενδεχομένω αρχίζει να τονώνει περισσότερο και την εσωτερική ζήτηση. Επιτέλου λοιπόν θα υπάρξει μια κάποια σύγκληση επειδή αυτή τη στιγμή προσπαθούμε να μειώσουμε το κόστος εργασίας και από την άλλη όμως προσπαθούμε να αυξήσουμε την παραγωγικότητα. Τώρα, πού βρίσκεται η Γερμανία αυτή τη στιγμή. Βρισκόταν στο 7% και παραμένει στο 7%. Ο τρέχον όμως λογαριασμός της Γερμανίας αυτή τη στιγμή δεν επιβαρύνει πλέον τις υπόλοιπες χώρες της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά επηρεάζει βέβαια και τον υπόλοιπο κόσμο. Πολλοί λένε ότι θα μπορούσε η Γερμανία να καταβάλει περισσότερε προσπάθειε προκειμένου να μην είναι επώδυνη προσαρμογή για τι υπόλοιπε χώρε. Ναι, ενδεχομένω ναι. Θα μπορούσαν να γίνουν κάποιε διορθώσει, αλλά αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι αρχίζεται αρχίζουμε να διορθώνουμε μια κατάσταση η οποία δεν ήταν βιώσιμη όλα αυτά τα χρόνια. Αρχίζει να διορθώνεται η κατάσταση αυτή και βλέπουμε τα, πρώτα θετικά αποτελέσματα. Η Ελλάδα αρχίζει και παρουσιάζει πλεόνασμα όσον αφορά τον προπολογισμό της και βλέπουμε ότι όλε οι χώρε αυτέ οι οποίε αναφερθήκατε αρχίζουν και αυτέ με τη σειρά του να παρουσιάζουν σιγά σιγά ένα πλεόνασμα στον προπολογισμό του. Τώρα έχουμε σοβαρά προβλήματα χρόνου. Έχουμε άλλε τέσσερι ερωτήσει. Ε, θα τι πάρουμε όλε μαζί. Και αν δεν ε, τελειώσετε εγκαίρω, ε, δεν θα προλάβετε να δώσετε συνέντευξη τύπου. Εσεί διαλέγετε. Μα είναι πιο σημαντικό αυτό από τη συνέντευξη τύπου, όντω, αλλά. Νομίζω ότι θα χρειαστούμε άλλη μισή ώρα να τα πάρουμε ξεχωριστά. Βέν Λάγκε, Ανκόκ, Μπόκροφ και Φιλίπ Λάμπρε. Ε, νόμιζα ότι θα είχαμε χρόνο και δέχτηκα και κάτι στη Τι να κάνουμε. Yeah. Ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Γενική Γραμματέα. Αν κλείσει το στόμα του ο δεν θα γίνουν καλύτερα τα πράγματα. Νομίζω πως η περιγραφή που κάνατε στο τέλος ότι οι εξαγωγές Γερμανίας δεν πάνε μόνο στην Ευρωζώνη αλλά πολύ πιο πέρα, ειδικά στην Ασία δεν θα αλλάξει τίποτα στις ανισότητες στην Ευρώπη. Τώρα εγώ έχω μια τελείως διαφορετική ερώτηση. Εδώ και 20 χρόνια εμένα με ενοχλεί το ότι ο ΩΣΑ δεν αναγνωρίζει την αξία της επαγγελματικής κατάρτισης. Ε, τα πιστοποιητικά επαγγελματικής κατάρτισης της Γερμανίας, εγώ θα έλεγα πως είναι εισάξια τουλάχιστον ε, με πτυχία ΤΕΙ, θα λέγαμε ή ε, κάποιο επίπεδο bachelor, κάτι το οποίο αρνείται ο ΣΑ να αναγνωρίσει. Αν δείτε όμως την ανεργία των νέων, πρέπει και ο ΩΣΑ κάποια στιγμή να δει την ιδέα πως δεν μπορεί να είναι τόσο λάθος αυτό το σύστημα της διπλής εκπαίδευσης σχολείου και επιχείρησης. Και το ερώτημά μου είναι, το σκέφτεται ο ο το ζήτημα, ίσως με τον ε, κύριο Λετέρν που γνωρίζει τα του καπιταλισμού του Ρήνου, όπως λέγεται. Να δείτε το σύστημα αυτό όταν υπάρχει 50% ανεργία των ε, νέων στην Νότια Ευρώπη και στην Γερμανία είναι μόλις 6,9%. Θα ακούσουμε όλες τις ερωτήσεις, οπότε θα απαντήσετε μία και καλή στο τέλος. Λοιπόν, Λία. Καλημέρα. Είμαι συνεισηγητής για την Τρόικα. Ε, αν πάω σε ένα, μια χώρα προγράμματος και του πω ότι είναι υπερβολική η αύξηση του μισθού σε σχέση με την παραγωγικότητα, δεν θα μάθει να πάρω καν το αεροπλάνο να γυρίσω κατά τη γνώμη μου. Τέλος πάντων, ε, σε σχέση με το υπερβολικό μοναδίο κόστος εργασίας συμφωνώ, αλλά βάσει του όσα πάλι ε, δεν αυξήθηκε ε, λόγω της αύξησης της κοινωνικής ασφάλισης, της αξίας κοινωνικής ασφάλισης, αλλά διότι είναι χαμηλότερη η ζήτηση σε αυτές τις χώρες. Οπότε εφόσον δεν πολλούνται τόσο πολλά εμπορεύματα, ο λόγος της παραγωγικότητας επί της απασχόλησης και άρα και το μοναδίο κόστος εργασίας εργασίας μειώθηκε και λοιπόν ε, αυτό εξηγεί τις αλλαγές στο μοναδιαίο κόστος εργασίας, ε, την αύξησή του δηλαδή. Το πρόβλημα δεν είναι η προσφορά, το πρόβλημα είναι η ζήτηση. Αυτό το συνεκτιμήσατε στους υπολογισμούς που κάνατε. Ευχαριστώ, Λες Μπρόκος. Ε, Ευχαριστώ. Θα ήθελα σας κάνω μία ερώτηση ε, για τα φορολογικά ζητήματα. Τέσσερα είναι οι βασικοί παράγοντες κατά τη γνώμη μου για τα φορολογικά ζητήματα. Ε, το δημοσιονομικό έλλειμμα, το δημόσιο χρέος, αλλά και ο ρόλος και η δομή του φορολογικού συστήματος. Ε, Εξού και η ερώτησή μου. Ποιες είναι οι πλέον σημαντικές φορολογικές μεταρρυθμίσεις που θα έπρεπε να γίνουν με τρόπο ώστε να συρρυκνωθεί ο φορολογικός τομέας κυρίως ε, στις νότιες χώρες και για να αναβαθμιστεί ε, το φορολογικό σύστημα πάλι στις ίδιες χώρες. Ε, πρόεδρος και τέλος, ο Φιλίπ. Καλώς ήρθατε κύριε Γκουρία. Συμφωνώ με πολλά πράγματα που είπατε για τη μεταρρύθμιση των τραπεζών, την ανάγκη να ασχοληθούμε με τη διαφύγη κτλ. Εσείς ζητήσατε ε, γρήγορα τον εύκολο στόχο που είναι η Διατλαντική Συμφωνία Εμπορίου, αλλά ο βασικός στόχος είναι να μειωθούν τα λεγόμενα μη δασμολογικά εμπόδια στο εμπόριο που συνήθως όμως ε, είναι περιβαλλοντικοί κανόνες, ε, υγειονομικοί κανόνες και κοινωνικοί. Δεν βλέπετε λοιπόν εδώ πέρα κάποιον κίνδυνο με το να επιδιώκουμε δηλαδή την κατάργηση των μη δασμολογικών εμποδίων στο εμπόριο, να αυξηθεί η πίεση της ανισότητας στην κοινωνία. Επανερχόμαστε στην αρχή λοιπόν και στο ερώτημα του Βέρνερ. Κοιτάξτε, δεξιότητες, δεξιότητες και πάλι δεξιότητες. Εγώ δεν συμφωνώ μαζί σας κύριε πως ο ΣΑ δεν ε, αξιολογεί την επαγγελματική κατάρτιση. Εμείς προσπαθούμε να πούμε πως έχει τόσο μεγάλη σημασία. Αλλά το πρόβλημα είναι πως εάν δεν ολοκληρωθεί ένας κύκλος δεν, και δεν πάρεις δίπλωμα δεν έχεις τίποτα στο τέλος. Προσπαθούμε να πούμε το εξή. Αν κάνεις ένα χρόνο, έχει ένα πιστοποιητικό ενός χρόνου, δύο χρόνια ένα πιστοποιητικό δύο ετών κτλ. Και αυτό κάτι αξίζει στην αγορά. Πρέπει να αλλάξει λίγο η νοοτροπία. Ότι εάν δεν τελειώσεις, δηλαδή, δεν έχει τίποτα στα χέρια σου. Γιατί πολλοί κόσμοι το εγκαταλείψει. Με δεύτερον, δεν μπορούν όλοι να πάνε στο πανεπιστήμιο, αλλά όλοι μπορεί να γίνουν ειδικοί μέσω της ε, επαγγελματική ε, κατάρτισης και οπωσδήποτε μετρήσαμε, όπως είπα, για πρώτη φορά 24 χώρες ε, ως προς τις δεξιότητες και λέμε ακριβώς πως δεν είναι μόνο η εκπαίδευση το ζήτημα, αλλά το πώς αυτή μεταφράζεται σε ικανότητες και δεξιότητες για να έχουν κάποια αξία οι άνθρωποι στην αγορά εργασίας. Ποια αγορά εργασίας. Όχι αυτή για την οποία τις προετοιμάζουμε, αλλά αυτή ε, που χρειάζεται στον πραγματικό κόσμο. Γιατί, Γιατί εδώ πέρα υπάρχει αναντιστοιχία. Παράγουμε ανθρώπους οι δεξιότητες των οποίων δεν χρειάζονται. Και υπάρχει παράδοξο. Εκατομμύρια ε, άνθρωποι άνεργοι, χιλιάδες εταιρείες ψάχνουν εργαζόμενους και δεν ε, τους βρίσκουν. Κάποιοι μάλιστα αναγκάζουν να φέρουν ανθρώπους από άλλες χώρες. Για μας λοιπόν το σύστημα αυτό το διπλό της εκπαίδευσης, η Γερμανία αυτή τη στιγμή ε, έχει τουρισμό από αυτή την υπόθεση, γιατί πάνε όλοι να δουν τι κάνει με την αγορά εργασίας, επειδή είναι τόσο επιτυχής. Και το ζήτημα του, της κουλτούρας αυτής μεταξύ ιδιωτικού τομέα συνδικάτων ε, και το πώς περνάνε σε part-time εργασία αντί να απολύουν κόσμο είναι πλέον μοντέλο. Οπότε προσπαθούμε να διαδώσουμε αυτές τις πρακτικές για το μοναδίο κόστο εργασία. Δεν είναι ζήτημα προσφοράς και ζήτησης. Ε, αναγνωρίζουμε ότι είναι χαμηλή η ζήτηση. Γιατί, γιατί η ανάπτυξη είναι χαμηλή. Ε, παντού αυτό. Εάν ε, ε είναι ανοιχτό το μαγαζί και πουλάει τα πάντα αλλά κανείς δεν αγοράζει, ε, τι να κάνουμε. είναι χαμηλή και η ανάπτυξη αυτό. Όμως δεν σημαίνει ότι απαραίτητα επηρεάζεται το, το κόστος εργασίας. Το θέμα είναι ότι χρειάζεται προσαρμογή διότι η παραγωγικότητα είναι μετρήσιμη. Κάθε μισά όρο, κάθε ώρα εργασίας τι παράγεται. Μπορούμε να το μετρήσουμε αυτό και αν ε, ε, την τελευταία δεκαετία, δεκαπενταετία έχουν αυξηθεί οι μισθοί περισσότερο σε σχέση με ε, τα προϊόντα, σε αυτά που έχουν παραχθεί, φυσικά δεν είμαστε ανταγωνιστικοί. Δεν έχει σχέση με την κρίση. Το πρόβλημα δεν είναι μόνο το ορεινό, δεν πρόκειται για τους προηγούμενους 18, τους επόμενους 18 μήνες, τα τελευταία 15 χρόνια. Και γι' αυτό ε, κάνουμε τις προτάσεις που κάνουμε. Να, μια, αυτό το, αυτή η γραφική αναπαράσταση είναι μια μικρή ιστορία, σύντομη ιστορία της ευρωπαϊκής οικονομίας. Εξηγεί ε, ε, σε μεγάλο βαθμό αυτά που συμβαίνουν σήμερα και βγαίνουν κάποιες εφημερίδες τώρα και τα κάνουν όλα περίπλοκα. Απλά είναι τα πράγματα, δείτε αυτό. Ε, ο δημόσιος τομέας ή μιλάτε για το φορολογικό τομέα. Θα έλεγα ε, πως δεν χρειάζεται να είναι ε, ιδίου μεγέθους όλες οι κυβερνήσεις γιατί δεν έχουν τις ίδιες ανάγκες. Όμως, παντού υπάρχουν δυνατότητες ε, μείωσης του κόστους, αλλά κυρίως παντού υπάρχει δυνατότητα παροχής αποτελεσματικότερων υπηρεσιών με χαμηλότερο κόστος. οι κρατικές επιχειρήσεις, χωρίς να με μπαίνουμε σε θρησκευτικά ζητήματα απελευθέρωσης κτλ. Σας μιλώ για ισότιμους όρους ανταγωνισμού. Το ζήτημα ε, της αρμοδιότητας της επιβολής φορολογίας, ε, γιατί ε, άλλο το θέμα της ίσπραξης των φόρων Με τη για την αρμοδιότητα επιβολής φόρων. Σχετίζεται άμεσα με τις δημόσιες υπηρεσίες. Παράδειγμα, τομέας υγείας. Εκεί σε όλες σχεδόν τις χώρες έχουμε τις υψηλότερες δαπάνες κατά κεφαλή. Ε, και ε, ταυτόχρονα εκεί σημειώνονται οι μεγαλύτερες αυξήσεις. Αυτό συνιστά πάρα πολύ μεγάλη απειλή. Θα δημιουργηθεί πάρα πολύ μεγάλο φορολογικό ζήτημα γιατί η γύρανση του πληθυσμού έρχεται να συνδυαστεί με την αύξηση των δαπανών στον τομέα της ε, υγείας και αυτό είναι θανατηφόρο για τους ε, κρατικούς προϋπολογισμούς ε, διότι η περίθαλψη που χρειάζεται για το γυράσκον πληθυσμό, για τις χρόνιες ε, παθήσεις ε, και ούτω καθεξής ε, επισύρουν μεγάλες δαπάνες. Λόγω της κρίσης δεν πρέπει μόνο να εξετάζουμε αν μπορούμε να τα καταφέρουμε καλύτερα. Εντάξει, ναι και αυτό. Ε, χρησιμοποιούμε αρκετά γενώσιμα. Ε, ελέγχουμε τις τιμές για τις φαρμακοβιομηχανίες, για την παραγωγή των φαρμάκων. Έχουμε ένα ε, ε, σύστημα ε, νοσοκομιακής περίθαλψης όπου πραγματικά ασχολούμαστε με αυτούς που χρειάζονται την νοσηλεία πραγματικά και όχι με αυτούς που θέλουν να γλιτώσουν τα ιατρικά έξοδα και νοσηλεύονται γι' αυτό. Υπάρχει το θέμα της πρόσβασης, της ποιότητας και του κόστους. Αυτό το ζήτημα ισχύει, αυτά τα ζητήματα ισχύουν και σε άλλους τομείς ίδρευση, ε, ε, αποχέτευση, οποιοδήποτε σύστημα και να πάρετε τα ίδια ισχύουν. Χρειαζόμαστε ε, ποιοτικέ, καλύτερε υπηρεσίε με χαμηλότερο κόστος. Γιατί, τι να σα πω, το σλόγγαν σήμερα είναι δημοσιονομική λιτότητα, σφιχτή προπολογισμή. Κύριε Λάμπρεχτ, Δεν είπα ότι είναι εύκολο το TTIP. Είπα η trade facilitation, η διατάξη περί διευκόλυνση των εμπορικών συναλλαγών στο Μπάλι είναι το, το πιο εύκολο, το πιο άμεσο που μπορούμε να επιτύχουμε, όχι η TTIP. Ε, και ακριβώς για τους λόγους που αναφέρατε κι εσείς. Υπάρχουν μη δασμολογικά ε, εμπόδια. Πρέπει να σας πω ότι σήμερα οι δασμοί που κυμαίνονται στο 3, 4, 5% δεν μας δίνουν έσοδα. Και άρα ε, ο παλιός τρόπος διαπραγμάτευσης τι ήταν. Εσείς θα μειώσετε τους δασμούς για τις τηλεοράσεις ε, και εμείς θα μειώσουμε ε, τους δασμούς για οτιδήποτε. Σε αντάλλαγμα για τα αυτοκίνητα ας πούμε. Έτσι διαπραγματευόμασταν παλιά. Σήμερα ξέρουμε ότι το καλύτερο που έχουμε να κάνουμε είναι μονομερής αφοπλισμός. Τι σημαίνει αυτό. Ε, ξέρουμε ότι η νέα βιομηχανική οργάνωση στον κόσμο είναι μια παραγωγή αλυσίδας αξιών, παγκόσμιας αλυσίδας αξιών. Τι σημαίνει όλο αυτό. Σημαίνει ότι μπορούμε να παράξουμε, είτε μιλάμε για τη Ρουάντα, είτε μιλάμε για την ε, Γερμανία, ένα κομμάτι αυτής της αλυσίδας αξίας με υψηλή εξειδίκευση. 40% ε, ε, των εξαγωγών ε, της αυτοκινητοβιομηχανίας της Γερμανίας, των μεγάλων βιομηχανιών, έχουν περιεχόμενο που δεν είναι γερμανικό. 50% των εξαγωγών των χωρών της G8 είναι υπηρεσίες. Και μια χώρα όπως η Γερμανία έχει μια πελώρια ανταγωνιστικότητα στη μεταποίηση πολιτική, αλλά χαμηλότατη στις υπηρεσίες. Για να διατηρηθεί λοιπόν στη ε, μεταποιητική η ανταγωνιστικότητα θα πρέπει να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα και στις υπηρεσίες. Αυτά δεν τα ξέραμε παλιά. Ε, η υπεραξία, η κινέζικη σε σχέση με τους Αμερικανούς, αν πάρουμε τη, ε, τους σχετικούς αριθμούς προστιθέμενης αξίας και όχι τους απόλυτους αριθμούς, ε, βλέπουμε μεγάλη μείωση στα ποσά με τα οποία κάνουμε τους υπολογισμούς μας. Αυτά τώρα τα ανακαλύψαμε μετά από μια απελώρια στατιστική και αναλυτική δουλειά που έχουμε κάνει ε, και αποκαλύπτονται αυτά. Δεν ήταν δυνατόν να τα ισχυριστεί αυτά κανείς ε, νωρίτερα σήμερα ή μάλλον το πάρουμε ανάποδα. Για να, ο καλύτερος τρόπος για να ε, εξασφαλίσουμε ανταγωνιστικότες σε εξαγωγές ε, είναι να, να βγάλουμε λίγο βάρος από τις ε, εισαγωγές. Ε, ο άλλος τρόπος είναι να είναι ακριβότερες οι εξαγωγές. μόνο έτσι μπορούμε μεταγενέστερα να καλύψουμε τις εμπορικές συναλλαγές. Σήμερα όμως δεν είναι δυνατόν να συμφωνήσουμε ήδη από σήμερα τι θα χρειαστούμε στο μέλλον να αφήσουμε την παπάγια να περιμένει στο λιμάνι μέχρι να σαπίσει. Ε, αυτό που χρειαζόμαστε είναι πληροφορίες ούτως ώστε να πηγαίνει το προϊόν στην αγορά που πρέπει τη στιγμή που πρέπει. Άλλη θεώρηση του παγκοσμίου εμπορίου χρειαζόμαστε και όχι τι μου δίνετε και τι σας δίνω, πάρε αυτό, δώσε αυτό. Και είναι αυτό σημαντικό γιατί το εμπόριο και πάλι θα είναι μεγάλη κινητήριος δύναμη της ανάπτυξης. Ε, thank and... Σας ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα όσα είπατε με τόσο ενθουσιασμό. Θεωρώ ότι ε, τα όσα κάνουμε εδώ στην Επιτροπή μας συνάδουν πάρα πολύ με αυτά τα οποία κάνετε και εσείς ε, στον ΩΣΑ και σε ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία δανείστηκα από τη δική σας την έκθεση και έβαλα στη δική μου. Θα ακούσουμε τώρα τον Επίτροπο Σέμετα και θα προεδρεύσει ο Πάμπλο γιατί εγώ πρέπει να συνοδεύσω τον κύριο Γκουρία σε μια συνέντευξη τύπου. Θα επιστρέψω πάντως. Ευχαριστώ Πάμπλο.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 Ας ξεκινήσουμε λοιπόν ευθύς αμέσως την ανταλλαγή απόψεων με τον κύριο Σεμέτα, Επίτροπο για τη Φορολογία και την Τελωνιακή Ένωση και την καταπολέμηση απάτης. Έχουμε λοιπόν ένα διαρθρωμένο διάλογο. Το πρώτο τμήμα θα έχει να κάνει με τις στατιστικές και το δεύτερο τμήμα θα έχει να κάνει με τη φορολογία. Θα ήθελα λοιπόν να δώσω καταρχάς για 10 λεπτά το λόγο στον Επίτροπο για να μας μιλήσει για τα στατιστική. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι εδώ στην Επιτροπή σας προκειμένου να κάνω μια σύντομη περίληψη των κοινών επιτευγμάτων μας. Μου δίνεται επίσης η δυνατότητα να αναφερθώ στα πιο σημαντικά νομοθετικά ζητήματα τα οποία αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα μπορέσω κατά αυτόν τον τρόπο να αναφερθώ και στο Ευρωπαϊκό Στατιστικό Σύστημα. Θα ήθελα να αναφερθώ καταρχάς σε κάποια συγκεκριμένα επιτεύγματα τα οποία απορρέουν από τη στενή συνεργασία που είχε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πρέπει να σας πω ότι το βελτιωμένο σύστημα επιτήρησης και συντονισμού όσον αφορά τα στατιστικά δεδομένα έχει προβλέψει πλέον νέες απαιτήσει σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο όσον αφορά την κατάρτιση στατιστικών δεδομένων. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να αρχίσουν να συγκεκριμένα μέτρα οικονομική πολιτική που θα κάνουν τα στατιστικά αυτά δεδομένα πιο αξιόπιστα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει πλέον πολύ πιο σημαντικά μέσα για να ελέγχει τα στατιστικά δεδομένα τα οποία παράγουν οι εθνικέ στατιστικέ αρχέ, καθώ επίση και τα δεδομένα αυτά τα οποία πορεύουν άμεσα από τι εθνικέ κυβερνήσει. Με κατεξοδότηση πράξη τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την οποία συνέβαλε πάρα πολύ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έχουμε πλέον πολύ συγκεκριμένε απαραίτητε λεπτομέρειε για τη διαδικασία διερεύνηση, ε, κακομεταχείρισης ή χειραγώγηση στατιστικών δεδομένων. Επίσης, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει καταφέρει να εντάξει στο six-pack, στην εξαπλή αυτή δέσμη οικονομικών μέτρων, συγκεκριμένες διατάξεις όσον αφορά την ανεξαρτησία και τον έλεγχο των εθνικών στατιστικών υπηρεσιών. Επίσης, υπάρχουν συγκεκριμένοι πλέον στατιστικοί δείκτες, οι οποίοι θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση των μακροοικονομικών ανισορροπιών. Όλα αυτά τα βήματα είναι πάρα πολύ σημαντικά για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ιδίω για την ε, Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Στατιστικών Δεδομένων, τη Eurostat, η οποία διαθέτει πλέον τα απαραίτητα μέσα. Κατά αυτόν τον τρόπο έχουμε βασικούς οικονομικούς δείκτες ύψης ποιότητα. Τα τελευταία γεγονότα καταδεικνύουν ότι δεν μπορούμε να έχουμε καμία εγγυημένη ποιότητα αν δεν υπάρχει απαραίτητος μηχανισμό ελέγχου είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε υψηλό επίπεδο διαφάνειας και λογοδοσίας. Αυτό ακριβώς προσπαθούμε να εντάξουμε στο Ευρωπαϊκό Στατιστικό Πρόγραμμα για το 2013, για την περίοδο 2013 μέχρι το 2017. Η επικοδομητική προσέγγιση της Επιτροπής Οικονομικής Πολιτικής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μας βοηθάει πλέον να έχουμε ένα πολύ καλό επίπεδο και ποιοτικά στατιστικά δεδομένα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Επίσης, καταφέρνουμε μέσω της ESA να έχουμε καλύτερα δεδομένα όσον αφορά τους εθνικούς λογαριασμούς. Θα πρέπει η ESA ε, να προσαρμοστεί προκειμένου να καταφέρουμε να, ε, να, ε, προκειμένου να ευθυγραμμιστεί περισσότερο με το Διεθνές Σύστημα Εθνικών Λογαριασμών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τα πιο σημαντικά ζητήματα. Όλα αυτά λοιπόν τα νομοθετήματα έχουν ολοκληρωθεί με επιτυχία και έχει ξεκινήσει και η εφαρμογή τους. Δεύτερον, θα ήθελα να αναφερθώ σε κάποια εκρεμή νομοθετήματα. Υπάρχουν ε, πολλές άλλες πρωτοβουλίες οι οποίες πρέπει να ολοκληρωθούν και γι' αυτό το λόγο χρειαζόμαστε τη δική σας την προσοχή και θα πρέπει να δράσετε αρκετά γρήγορα. Αναφίβολα το πιο σημαντικό τέτοιο νομοθέτημα είναι ο λεγόμενος statistical law, το νομοσχέδιο δηλαδή για, την, για τα στατιστικά δεδομένα. Θεωρώ ότι είναι το πιο σημαντικό νομοθέτημα που αφορά τόσο το Eurostat όσο και τις Εθνικές Υπηρεσίες Στατιστικών Δεδομένων. Από το 2011 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει ζητήσει τα απαραίτητα εχέγγυα για την αξιοπιστία των ευρωπαϊκών στατιστικών, ιδίω στα πλαίσια μια ε, βελτιωμένη οικονομική διακυβέρνηση. Η πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την αθεώρηση του στατιστικού νόμου μου δικαιολογείται ακριβώ για τι ίδιε αρχέ. Θα πρέπει να καταφέρουμε να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα που έχουν ε, εντοπιστεί σε ορισμένα κράτη-μέλη. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταφέρουμε στα πλαίσια τη οικονομική κρίση να βελτιώσουμε το πρόβλημα αξιοπιστία που υπάρχει με ορισμένα ευρωπαϊκά στατιστικά δεδομένα. Θα πρέπει καταρχά να εγγυηθούμε την επαγγελματική ανεξαρτησία των εθνικών στατιστικών υπηρεσιών και κατά δεύτερο λόγο θα πρέπει να έχουμε ένα στατιστικό συντονισμό σε εθνικό επίπεδο. Πέρυσι το Δεκέμβριο η Επιτροπή ΕΚΟΝ σχεδόν ομόφωνα ενέκρινε ένα σχέδιο έκθεσης που ακολουθεί τη λογική αυτή. Αυτό που μας ανησυχεί όμως είναι ότι ε, όλες ε, οι προτεραιότητες αυτή τη στιγμή έχουν μετακινηθεί περισσότερο προς τον σχεδιασμό της Eurostat και όχι τόσο πολύ στο να εξευρεθούν κάποιες πραγματικές λύσεις για τον τρόπο που λειτουργούν τα εθνικά συστήματα, οι εθνικές υπηρεσίες στατιστικών δεδομένων. Έχουμε πλέον την πλήρη ανεξαρτησία της ε, Eurostat και η εμπειρία που έχουμε μέχρι στιγμής καταδεικνύει ότι ε, η Eurostat ανταποκρίνεται στις αρμοδιότητές της και στις προσδοκίες σας. Αυτό άλλωστε έχει επιβεβαιωθεί από τις εκθέσεις ε, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για την Στατιστική Διακυβέρνηση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση όμω από μόνη τη δεν μπορεί να εγγυηθεί την αξιοπιστία των ευρωπαϊκών στατιστικών δεδομένων. Εξαρτώμεθα πάρα πολύ από την αξιοπιστία των δεδομένων που φτάνουν από τις Εθνικές Στατιστικές Υπηρεσίες. Τα πρότυπα λοιπόν θα πρέπει να είναι κοινά σε όλα τα επίπεδα παντού στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Ευρωπαϊκό Συμβουλευτικό Όργανο για τις ε, Στατιστικές ακριβώς τι ανησυχίες έχει εκφράσει στην ετήσια έκθεσή του του 2013 που πρόσφατα κατατέθηκε και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Επίσης, έχουμε κάποιες ε, διατάξεις όσον αφορά τον Γενικό Διευθυντή της Eurostat που δεν σέβονται την θεσμική ισορροπία που έχουμε στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πολλές φορές διατάξεις που προβλέπονται επίσης έχουν δημιουργήσει μια ανισορροπία στις σχέσεις της Eurostat με τις εθνικές στατιστικές υπηρεσίες. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταφέρουμε σε αυτή τη στρατηγική μεταρρύθμιση να πετύχουμε την κατάλληλη ισορροπία. Ήδη αρχίσαμε να επεξεργόμαστε την πρόταση για έναν κανονισμό παροχής ποιοτικών στατιστικών δεδομένων όσον αφορά την διαδικασία μακροοικονομικής ανισορροπίας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε ποιοτικά στατιστικά δεδομένα που θα μας επιτρέπουν να αξιολογούμε σωστά την όλη διαδικασία μακροοικονομικής ανισορροπίας. Αυτό άλλωστε έχει ζητήσει ήδη από τον Νοέμβριο του 2011 το Συμβούλιο ΕΚΟΦΗΝ. Χαιρετίζουμε το σχέδιο έκθεσης του κυρίου Έπινγκ και όλους ιδιαίτερους η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χαιρετίζει το γεγονός ότι ο εισηγητής υποστηρίζει την ε, ανάγκη να βελτιωθεί το σύστημα επιτήρησης των στατικών δεδομένων όσον αφορά τη διαδικασία μακροοικονομικής ανισορροπίας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να εντοπίζονται συγκεκριμένες διαδικασίες για την αξιολόγηση της ε, διαδικασίας μακροοικονομικής ανισορροπίας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να επιτύχει, να κλείσει το φάκελο αυτό το συντομότερο δυνατό και στηρίζομαι στην υποστήριξη και την κατανόηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το στόχο αυτό. Τρίτον, ολοκληρώνοντα την παρέμβασή μου αυτή, θα ήθελα να αναφερθώ σε κάποια συγκεκριμένα σχέδια όσον αφορά κάποιου βασικού στατιστικού δείκτε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Sharon Bowles για τον επικοδομητικό ρόλο που έχει διδραματίσει, ιδίω στα πλαίσια τη διάσκεψη για την εφαρμογή του ΕΨΑΣ, δηλαδή των ευρωπαϊκών προτύπων όσον αφορά τα δημόσια στατιστικά δεδομένα. Η διάσκεψη αυτή έλαβε χώρα τον Μάιο του 2013 και καταδεικνύει η διάσκεψη αυτή ότι πραγματικά πρέπει να καταλήξουμε αυτή τη στιγμή σε κάποιου εναρμονισμένους κανόνες όσον αφορά τα δημόσια στατιστικά δεδομένα. Χάρη στο ΕΨΑΣ θα έχουμε μεγαλύτερη συγκρισιμότητα των χρηματοοικονομικών δεδομένων και κατά αυτόν τον τρόπο και καλύτερο οικονομικό συντονισμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα καταφέρουμε να βελτιώσουμε επίση την χρηματοοικονομική διαχείριση όλων των κυβερνητικών φορέων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα προωθήσει λοιπόν το σχέδιο αυτό χάρη στην πολύ καλή υποστήριξη που έχει μέχρι Το επόμενο στάδιο θα είναι να εντοπίσουμε και να προτείνουμε τις βασικές αρχές του σχεδίου αυτού, καθώς επίσης και έναν συγκεκριμένο χάρτη πορείας για την έγκρισή του. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσβλέπει στην ισχυρή υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προκειμένου το σχέδιο έψας τελικά να καταρτιστεί και να εφαρμοστεί. Μια άλλη σημαντική πρωτοβουλία για το Ευρωπαϊκό στατιστικό σύστημα είναι να υπάρχει ένας νέος γύρος εκθέσεις ομοτήμων όσον αφορά τις βασικές αρχές του κώδικα δεοντολογίας για τις ευρωπαϊκές στατιστικές. Σύμφωνα με τις συστάσεις που έχει κάνει το Ευρωπαϊκό Συμβουλευτικό Όργανο για, τις, για τα στατιστικά δεδομένα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, υποβάλλονται συγκεκριμένε προτάσεις συντονισμού προς τις Εθνικές Υπηρεσίες Στατιστικών δεδομένων προς τις Εθνικές Στατιστικές Υπηρεσίες. Ένα πιλωτικό πρόγραμμα ήδη έχει ολοκληρωθεί και θα καταφέρουμε να πετύχουμε κατά αυτόν τον τρόπο μια μεγαλύτερη συμμόρφωση όλων των εθνικών στατιστικών υπηρεσιών με τον Ευρωπαϊκό Κώδικα Δεοντολογίας. Κατά αυτόν τον τρόπο θα καταφέρουμε να πετύχουμε ένα πιο βελτιωμένο και ποιοτικό σύστημα Στατιστική διακυβέρνηση, τόσο σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση, όσο και σε εθνικό επίπεδο. Τέλο, να σα πω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ξεκινήσει μία ει ανάλυση προκειμένου να εξυγχρονιστεί ο τρόπος παραγωγής ευρωπαϊκών στατιστικών και να εξυγχρονιστεί επίσης και η διακυβέρνηση των ευρωπαϊκών στατιστικών. Το σχέδιο αυτό έχει ξεκινήσει από την Eurostat καθώς επίσης και από του εταίρους της Eurostat στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Στατιστικής. Πολλά κράτη-μέλη έχουν αρχίσει να συμμετέχουν σε μια ομάδα υψηλού επίπεδου θα αποτελέσει η εργασία της ομάδας αυτής εργασίας μια πρώτη βάση προκειμένου να καταφέρουμε τον Μάιο του 2014 να έχουμε μια πιο ευρεία συζήτηση στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του Στατιστικού Συστήματος. Καταλαβαίνετε λοιπόν ποιε είναι οι προκλήσει που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσον αφορά τα ευρωπαϊκά στατιστικά δεδομένα. Καλούμε θα ανταποκριθούμε στι προκλήσει αυτέ με τον πιο αποδοτικό τρόπο. Ξέρετε ότι πρέπει να γίνουν σημαντικέ οικονομικέ και διοικητικέ προσπάθειες είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει πολιτική υποστήριξη σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο και συνεχίζω να ελπίζω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα συνεχίσει να μας υποστηρίζει προκειμένου να καταφέρουμε να καταστήσουμε τις ευρωπαϊκές στατιστικές πιο αξιόπιστες και πιο χρήσιμες. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Σεμέτα. Θα δώσω πρώτα απ' όλα τον λόγο στον συντονιστή του ΕΛΚ, τον κύριο Γκοζές και μετά θα απαντήσετε. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ κύριε Επίτροπε που ήρθατε για μια φορά ακόμα για να μας κάνετε παρουσίαση εδώ στην Επιτροπή μας. Θα ήθελα να κάνω δύο συγκεκριμένες ε, ερωτήσεις. Καταλαβαίνω ότι σε μεταγενέστερο στάδιο θα καταφέρετε να μου δώσετε πιο συγκεκριμένη απάντηση. Πάντως θα ήθελα να εκφράσω δύο ανησυχίες που έχω αυτή τη στιγμή, ιδίως όσον αφορά τη Γαλλία. Θα ήθελα να γνωρίζω καταρχάς αν έχει ληφθεί μία μια απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσον αφορά τον χαμηλό φόρο προστιθέμενης αξίας για τα ψηφιακά βιβλία στην Γαλλία, αν έχετε αναλύσει το ζήτημα αυτό και αν έχετε καταλήξει σε κάποια απόφαση. Και η δεύτερη ερώτησή μου έχει να κάνει πάλι με το φόρο προστιθέμενης αξίας. Ξέρετε ότι ε, την Κυριακή αυτή στην Γαλλία είχαμε πάρα πολλές διαδηλώσεις και είχαμε πάρα πολλά άλογα στους ε, δρόμους των γαλλικών πόλεων, πάλι επειδή προβλέπεται μία αύξηση του φόρου προστιθέμενης αξίας όσον αφορά τα άλογα αυτή τη φορά. Ξέρετε ότι κατηγορούμε πάρα πολύ συχνά την Ευρωπαϊκή Ένωση για την αύξηση του φόρου προστιθέμενης αξίας στις δύο αυτές κατηγορίες, από την άλλη όμως φαίνεται ότι τα πράγματα είναι αρκετά πολύπλοκα και ότι ενδεχομένως θα μπορούσαμε τουλάχιστον να έχουμε μειωμένο φόρο τη θέμενη αξίας όσον αφορά κάποιους συγκεκριμένου τομεί. Ότι θα μπορούσε να γίνει μια εξαίρεση όσον αφορά τα στοιχήματα ή όσον αφορά την αγοροπολισία αλόγων που συμμετέχουν σε αγώνες. Ξέρετε ότι είναι συγκεκριμένε πληροφορίε που φτάνουν αυτή τη στιγμή προ τον Γάλλο ψηφοφόρο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό οι Γάλλοι ψηφοφόροι να γνωρίζουν ακριβώ ποια είναι η άποψη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γιατί ξέρετε ότι πολλέ φορέ η σύγχυση αυτή χρησιμοποιείται από διάφορε ομάδε πολιτικέ που είναι κατά τη Ευρωπαϊκή Ένωση ξέρω αν έχετε ερωτήσει για τη φορολογία, δεν είναι ερώτηση για τη φορολογία. Αυτό δεν ξέρω αν θέλετε να απαντήσετε κύριε Επιτροπέ. Ναι βεβαίω. Υποτίθεται ότι θα μιλούσαμε για στατιστικά στοιχεία, αλλά η ερώτηση αυτή αφορά τη φορολογία. Σημαντικό θέμα να απαντήσω. Όσον αφορά το μειωμένο ΦΠΑ. Ξέρετε πως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεσμεύτηκε για να κάνει μια αξιολόγηση του συστήματος μειωμένου ΦΠΑ. Η αξιολόγηση αυτή συνεχίζεται. Τελείωσε η δημόσια διαβούλευση. Έχουμε ζητήσει και δύο μελέτες αξιολόγησης και αυτή τη στιγμή οι υπηρεσίες μου εξετάζουν την αξιολόγηση αντικτύπου που θα ολοκληρωθεί στο τέλος του έτους, αρχές του επόμενου έτους. Και αυτή η αξιολόγηση θα δημοσιευτεί σε όλους τους ενδιαφερόμενους. Δεύτερο ζήτημα που αφορά τον ΦΠΑ ε, στα άλογα και στις σχετικές υπηρεσίες. Υπάρχει εδώ πέρα μία απόφαση του ελεκτικού, όχι με συγχωρείτε, του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, για το ότι ο μειωμένος ΦΠΑ που ίσχυε για το θέμα αυτό στη Γαλλία αντίθετος ε, με την οδηγία του ΦΠΑ. Και μια που επικρατεί βεβαίως ε, ένα σύστημα κράτους δικαίου, όλα τα κράτη-μέλη και η Γαλλία πρέπει να εφαρμόσουν αυτό το οποίο τα ίδια τα κράτη ομόφωνα συμφώνησαν στο Συμβούλιο. Θα ήθελα να σας πενθυμίσω πως το 2009 όταν έγινε η τελευταία αναθεώρηση του ΦΠΑ και τότε είχαμε το θέμα του μειωμένου ΦΠΑ στην εστίαση η Γαλλία δεν έθεσε τότε το ζήτημα αυτό για τα άλογα. Και η οδηγία παραμένει ίδια. Άρα η Γαλλία, όπως και όλα τα κράτη-μέλη, πρέπει να εφαρμόσει τις διατάξεις ε, της οδηγίας που έχει συμφωνήσει. Δεν υπάρχουν άλλοι τρόποι για να βοηθήσετε τον κλάδο αυτόν και νομίζω πως και η γαλλική κυβέρνηση θα μπορούσε να εφαρμόσει κάποια μέτρα και μπορούν να χρησιμοποιηθούν και κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη στήριξη του κλάδου αυτού. Η Κομισιόν ε, είναι διατεθειμένη να συνεργαστεί με τις γαλλικές αρχές για να βρεθούν άλλοι τρόποι για να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα αυτού του κλάδου. Σας ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Ο κύριος ε, Αγγιόκ για τους ε, σοσιαλιστές. Ευχαριστώ Παύλο. Καλημέρα Επίτροπε. Χαίρομαι που μπορούμε να κάνουμε έναν απολογισμό μαζί, λίγες ημέρες μόνο, μετά την ψηφοφορία στο Κοινοβούλιο για την αναθεώρηση του κανονισμού για τις ε, ε, στατιστικές. Την ε, περασμένη Πέμπτη εγκρίθηκε ο κανονισμός με 617 ψήφους υπέρ και 20 κατά. Ενισχύεται η ανεξαρτησία και ε, η νομοποίηση των Εθνικών Στατιστικών Ιδρυμάτων με τον κώδικα διοντολογίας ε, ενισχύεται ε, η αρμοδιότητα, η διερευνητική αρμοδιότητα και η συντονιστική αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Στατιστικό Σύστημα. η βασική έρηδα με εσάς έγκυται στις προτάσεις που κάνουμε για τη Eurostat. Ε, κρίνουμε ότι είναι απαραίτητο να ενισχυθεί η ανεξαρτησία του Γενικού Διευθυντή και της Eurostat, όχι διότι τίθεται να αμφιβόλω σήμερα, αλλά για να αντιμετωπίσουμε τα, τους απρόβλεπτους παράγοντες. Είδαμε τι συνέβη με την ε, κρίση στην Ελλάδα, αν αυτά ίσχυαν τότε, τα όσα ισχύουν σήμερα ίσχυαν τότε, θα ήταν διαφορετική η κατάσταση. Επίσης, σε άλλο σημείο τριβής ήταν ο διορισμός του Διευθυντή της Eurostat θα πρέπει να εκφεύγει ε, ασδήποτε πολιτικής πίεσης ο διευθυντής ε, της Eurostat, ε, όμως με τις αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την οικονομική διακυβέρνηση έχει πολιτικό ρόλο πια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δείτε την επιρροή που έχει στην Τρόικα ή δείτε την επιρροή που έχει στη διαδικασία Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Δεν θέλουμε ε, άρδιν ε, να αναθεωρήσουμε την ε, ισορροπία δυνάμεων και να δημιουργήσουμε προηγούμενο που θα πλήξει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όχι, απλώς μιλάμε για την Eurostat την Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία. Θέλουμε μεγαλύτερη ανεξαρτησία και διαφάνεια για τα, ε, για τα εθνικά ε, στατιστικά ιδρύματα ε, και ε, θέλουμε να δίνει το παράδειγμα η Eurostat. Ε, Επίση, συμφωνούμε ως επιτοπλίστων με το Συμβούλιο για το μεγαλύτερο μέρος του κανονισμού. μέχρι στιγμής η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη διαφούλευση του Κοινοβουλίου δημιουργεί νέα εμπόδια. Σας ερωτώ πολύ απλά Προτίθεστε να συνεργαστείτε μαζί μας για να καταλήξουμε τελικά σε μια συμβαστική λύση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ερωτήσεις σας και καλημέρα. Επίσης. Ε, χαίρομαι που συνεχίζουμε τη συζήτηση μετά την ψηφοφορία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου επί του κανονισμού. Κάποια πράγματα είπατε στην παρέμβασή σας πως εάν υπήρχε ο κανονισμός πριν από τρία χρόνια, τέσσερα, πέντε, Ό,τι πιθανώς δεν θα είχαμε προβλήματα με τα ελληνικά στατιστικά στοιχεία. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο γιατί το πρόβλημα των ελληνικών στατιστικών στοιχείων ξεκίνησε με τα ηλεκτρονικά δεδομένα ήδη. Και από το 2005 υπήρχαν τροποποίησεις του κανονισμού για να αντιμετωπιστούν ε, τέτοια προβλήματα. Αλλά δυστυχώς τότε τα κράτη-μέλη δεν ήταν σε θέση να συμφωνήσουν στην ε, πρόταση. Φαίνεται πως ε, πράγματι είχαν ε, από τότε πρόβλημα τα ελληνικά στατιστικά στοιχεία. Τώρα η συμφωνία ενίσχυσε την Eurostat αλλά τώρα επετεύχθη η συμφωνία. Βεβαίως ο κοινό μας στόχος είναι να καταλήξουμε σε μια οριστική συμφωνία για το λεγόμενο στατιστικό δίκαιο και όπως είπα και στο Κοινοβούλιο, στην Ολομέλεια του Στρασβούργου, η Κομισιόν βεβαίως είναι διατεθειμένη να συζητήσει, να διαπραγματευτεί έναν συμβιβασμό και θα προσπαθήσει να κάνει ό,τι μπορεί για να συμβιβάσει τις θέσεις ε, Συμβουλίου και Κοινοβουλίου σε κάποια συγκεκριμένα ζητήματα. Και νομίζω είναι σημαντικό να έχουμε τον ίδιο στόχο, δηλαδή να ισχυροποιηθεί το Ευρωπαϊκό Στατιστικό Σύστημα και Ε, επί τη βάση αυτή νομίζω πως έχουμε κάποια ζητήματα να αντιμετωπίσουμε μεταξύ των οποίων και η Eurostat. Επίσης οφείλω να αναφερθώ στην ε, πρόσφατη έκθεση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για τα στατιστικά στοιχεία που έκανε μια ανεξάρτητη αξιολόγηση της Eurostat ε, και την έκθεση την έχετε στη διάθεσή σας ε, πως η Eurostat έχει πλήρη ανεξαρτησία και ανταποκρίνεται στις απαιτήσει ε, του κώδικα συμπεριφοράς. Σημαντική πληροφορία νομίζω που πρέπει να ληφθεί υπόψη όταν θα συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις πάνω στο σημαντικό αυτό θέμα. Αλλά όπως είπα θα καταβάλουμε κάθε προσπάθεια. Ήδη οι υπηρεσίες μου έχουν ξεκινήσει να αναζητούν ε, μια πιθανή ε, λύση στο θέμα αυτής της ε, νομοθεσίας. Σας ευχαριστώ για τους Ευρωπαίους συντηρητικούς και μεταρρυθμιστές. Ναι, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, σας ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια για την έκθεσή μου για την ποιότητα στατιστικών στοιχείων. Για την διαδικασία μακροοικονομικών ανισορροπιών. Η ερώτησή μου αφορά τον φόρο χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών που συζητήθηκε εδώ πέρα πριν από τρία χρόνια νομίζω πρώτη φορά που είπα πως ο φόρος αυτός είναι ένα εξαιρετικό παράδειγμα μιας κακής ιδέας. Πρόσφατα ε, κεντρική τράπεζα, ο κεντρικός τραπεζίτης της Γαλλίας είπε πως ε, απειλεί ο φόρος αυτός τη δημοσιονομική σταθερότητα. Επίσης, ένα μήνα μετά, η νομική υπηρεσία του Συμβουλίου είπε πως είναι παράνομος αυτός ο φόρος γιατί έχει εξοεδαφικότητα. Μετά η Bundesbank είπε πως ε, τα κράτη-μέλη θα εξαρτούν περισσότερο από φτηνά λεφτά της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Έχουμε λοιπόν εδώ πέρα ένα παράδειγμα φόρου που έχουμε ξοδέψει ήδη δύο φορές τα προσδοκόμενα έσοδα χωρίς να έχουμε εισπράξει ακόμα τίποτα. Δεδομένων όλων αυτών των προβλημάτων και των περιορισμένων πόρων σας, μήπως παταλάτε το χρόνο σας με τον φόρο αυτόν. Ευχαριστώ. Συζητήσαμε για τη φορολογία, λέει η πρόεδρος, αλλά αν θέλετε να απαντήσετε. Φαίνεται πως ε, είναι πιο ενδιαφέρουσες οι ερωτήσεις για τη φορολογία παρά για τα στατιστικά στοιχεία. Αν και εγώ θεωρώ πως είναι εξίσου σημαντικά. Λοιπόν, για το φόρο χρηματοοικονομικών συναλλαγών. Να σας υπενθυμίσω πως ε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με συντριπτική πλειοψηφία προσφάτως ε, υπερψήφισε την πρόταση για τον φόρο με κάποιες πολύ καλές ιδέες για το πώς μπορεί να βελτιωθεί η πρόταση αυτή και νομίζω πως τα κράτη-μέλη θα αναλύσουν ε, τις ιδέες αυτές που περιέχονται στην έκθεση του Κοινοβουλίου και δεν αμφιβάλλω πως κάποιες από αυτές θα υιοθετηθούν στις ε, διαπραγματεύσεις. Κατόπιν, πάρα πολλοί αναφέρθηκαν στη γνωμοδότηση της νομικής υπηρεσίας του Συμβουλίου. Και έβγαλαν κάποια γενικά συμπεράσματα. Θα ήθελα να επισημάνω πως η νομική υπηρεσία του Συμβουλίου γνωμοδότησε για πολύ συγκεκριμένα σημεία της πρότασης για τον φόρο αυτόν. Όχι για την πρόταση στο σύνολό της, αλλά για μία παράγραφο ενός άρθρου. Και η Κομισιόν θεωρεί πως η γνωμοδότηση αυτή δεν είναι σωστή. Η Δενομική Υπηρεσία της Κομισιόν ήδη έχει συντάξει μια έκθεση η οποία θα παρουσιάσει σαφή επιχειρήματα για το γιατί θεωρούμε λανθασμένη τη νομοδότηση αυτή και η έκθεση αυτή θα παρουσιαστεί στα κράτη-μέλη στην επόμενη συνεδρίαση της ομάδας εργασίας στις 12 Δεκεμβρίου. Και είμαστε πεπισμένοι πως η θέση της Κομισιόν στο ζήτημα αυτό ήταν η σωστή. Και πως η πρόταση ίδια σέβεται πλήρως ε, τις διατάξεις της συνθήκης. Κατόπιν, δεν πρέπει να ξεχνάμε πως με τον ε, φόρο αυτόν ε, είμαστε στη διαδικασία ενισχυμένης συνεργασίας. Αυτό σημαίνει πως 11 κράτη-μέλη εθελοντικά συμφώνησαν να προχωρήσουν στο θέμα αυτό και να βρουν ένα συμβιβασμό μεταξύ τους για το πώς θα εισαχθεί ο φόρος αυτός χρηματοοικονομικών υπηρεσιών στις 11 αυτές χώρες. Το θέμα λοιπόν τώρα είναι στα χέρια των κρατών μελών. Αναμένουμε την περαιτέρω πρόοδο. Ολοκληρώθηκε η πρώτη ανάγνωση στο Συμβούλιο και τώρα πρέπει να υπάρξει ένας πολιτικός συμβιβασμός και ελπίζω τα κράτη-μέλη που συμμετέχουν να έχουν την πολιτική βούληση για να συμφωνήσουν στον πολιτικό συμβιβασμό του των δυνατών. Ο Φιλίπ για τους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 Ευχαριστώ, Επίτροπε, για τις στατιστικές εργασίες. Ε, γνωρίζετε πόση σημασία προσδίδουμε στην επέκταση του σετ δικτών πέρα από το παραδοσιακό ΑΕΠ που χρησιμοποιούμε αδιακρίτως παντού και να ε, επεκτείνουμε λοιπόν το σετ δικτών στο περιβαλλοντικό τομέα, στο κοινωνικό τομέα. Σας ερωτώ λοιπόν, έχει σημειωθεί καμία πρόοδος ε, για αυτού του είδους τους δείκτες και πώς μπορεί να επηρεαστεί η διαδικασία λήψη αποφάσεων στην Ευρώπη με τη χρήση αυτών των δικτών Πώ ε, πώς θα προσδιορίσουμε τι χρειαζόμαστε και πώς θα συλλέξουμε στη συνέχεια τα στοιχεία που θα έχουμε προφασίσει. Απάντηση. Αληθεύει όπως πολύ καλά γνωρίζετε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πραγματεύεται αυτό το ζήτημα και έχουμε και ένα συγκεκριμένο σχέδιο υπέρ, πέραν του ΑΕΠ. Θα συμπεριλαμβάνεται λοιπόν δείκτης ε, θα συμπεριλαμβάνονται δείκτες ε, που σχετίζονται όχι μόνο με το ΑΕΠ, αλλά θα εξηγούν ποια είναι η επίπτωση του ΑΕΠ ε, σε διάφορες κοινωνικές πληθυσμιακές ομάδες, πώς επηρεάζεται η οικονομία και το καθεξής. Ο συνάδελφός μου θα μπορούσε ίσως να μας ενημερώσει για την ε, πρώτη δημοσίευση των στοιχείων ε, της μελέτης αυτής, γιατί είμαστε σε στενή συνεργασία και με τον ΟΣΑ για αυτό το ζήτημα. Κατά την ε, προσωπική μου άποψη, ένα από τα προβλήματα αυτού του σχεδίου είναι το κατά πόσο είναι επίκαιροι οι διάφοροι δείκτες. Υπάρχουν μεγάλες διαφοροποιήσεις, δηλαδή την στιγμή που είμαστε έτοιμοι να κοινοποιήσουμε τα στοιχεία του ΑΕΠ μετά την εκπνοή της ε, περίοδου αναφοράς. Άλλα στοιχεία δεν είναι ακόμη διαθέσιμα. Δεν μπορούμε ταυτόχρονα δηλαδή να κοινοποιήσουμε τους διαφόρους δείκτες ε, και ε, εξού και το πρόβλημα. Πώς μπορούμε να αμβλύνουμε αυτές τις διαφορές ε, ώστε ταυτόχρονα μπορούμε να δημοσιεύουμε στοιχεία που σχετίζονται με το ΑΕΠ και την επίπτωση, χάρη του, την επίπτωση της μείωσης του ΑΕΠ επί διαφόρων οικονομικών μεγεθών. Μπορείτε να επεκταθείτε εσείς παρακαλώ για αυτό το ζήτημα. Ε, σε σχέση με αυτά που είπε ο Επίτροπος Σεμέτα, έχουμε δύο διαφορετικές προσεγγίσεις. Η μία είναι να επεκτείνουμε το πεδίο ούτως ώστε να καλύψουμε τη, αυτά που, αυτό που καλούμε πρόοδο των κοινωνιών. Και μαζί με το ταχύμετρο που είναι το ΑΕΠ να έχουμε και ένα κατάλογο δικτών που ε, ε, καλύπτει ε, το διαθέσιμο εισόδημα των οικοκυριών, τα κοινωνικά και περιβαλλοντικά ζητήματα. Σε σχέση με τη δημοσίευση, τις επόμενες και προηγούμενες δημοσίευσεις, να σας πω ότι τον Οκτώβρη Έχουμε μια, είχαμε μια δημοσίευση για τους δείκτες ε, της Ευρώπης 2020. Δείξαμε όλη τη σειρά των δικτών σε σχέση με τις ε, ε, στοχευμένες αξίες που είχαν αποφασιστεί και σε ευρωπαϊκό και σε εθνικό επίπεδο. Τις επόμενες μέρες ή και εβδομάδες θα δημοσιεύσουμε την έκθεση παρακολούθησης για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Είναι μια διετής έκθεση που επίσης ε, προσμετρά όλους τους δείκτες με ευανάγνωστο εύληπτο τρόπο ή τουλάχιστον το ελπίζω. Η δεύτερη προσέγγιση είναι να επιταχύνουμε όπως είπε και ο Επίτροπος ε, σε τομείς όπου ε, από διαρθρωτικής πλευράς έχουμε χρονοκαθυστέρηση σε σχέση με την διαθεσιμότητα των στοιχείων αφενός στο ΕΠ και αφετέρου των κοινωνικοπεριβαλλοντικών στοιχείων. Δυστυχώς αυτό ισχύει για ολόκληρο το φάσμα των δικτών Εστιάζουμε την προσοχή μας όμως στο θέμα των αερίων του θερμοκηπίου, τα ενεργειακά ζητήματα και χρησιμοποιούμε ως ενδεικτικούς αυτούς τους δείκτες. Ε, και επίσης βάσει της ενεργειακής κατανάλωσης κάνουμε προβλέψεις για τα στοιχεία που θα έχουμε για το διοξίδιο του άνθρακα, προσεγγίζοντας έτσι στο μέτρο του δυνατού ε, αυτά τα στοιχεία με τα οικονομικά στοιχεία για ε, τους ε, κοινωνικούς όμω ε, όμως και τον επιμερισμό του πλούτου στα νοικοκυριά έχουμε μεγάλη καθυστέρηση και βλέπουμε ότι η κρίση έχει επηρεάσει σε τόσο μεγάλο βαθμό τα κράτη-μέλη που θα πρέπει να έχουμε περισσότερα στοιχεία σε σχέση με την φτώχεια, τις εισοδηματικές ανισότητες και τα λοιπά. Προσπαθούμε πάντως και φτάνουμε στο όριο των, του δυνατού για τους στατιστικολόγους. Ε, ευχαριστώ. Από την ΚΟΕ έχουμε ερωτήσεις. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θέλω να πω ότι η ερώτησή μου είναι για τη φορολογία. Βέβαια στη συνέχεια τα μπερδέψαμε τα θέματα. Δεν ξέρω αν υπάρξει δεύτερος γύρος για να μην ευθυνδιάσω τον Επίτροπο. Αλλά από ό,τι είδα γίνονται και τέτοιες ερωτήσεις, αν μου επιτρέπετε την κάνω. Δεν είναι για τα στατιστικά, κατάλαβα ότι ενδεχομένω θα έχουμε δύο γύρου. Λοιπόν, αν μου δίνετε την άδεια, κάνω την ερώτηση. Ευχαριστώ πολύ. Ναι, ναι, ευχαριστώ πολύ τον κύριο Επίτροπο που ευρίσκεται εδώ. Και με την ευκαιρία, η ερώτηση μου είναι πάρα πολύ ευαμπλή, κύριε Σεμέτα. Πριν δύο χρόνια είχα ρωτήσει την Κομισιόν αν ήταν ευχαριστημένη από την πάταξη της φοροδιαφυγής, της μεγάλης φοροδιαφυγής στην Ελλάδα. Πριν δύο χρόνια. Η απάντηση που είχε δώσει είναι ότι η πάταξη της φοροδιαφυγής είναι βασικό στοιχείο του προγράμματος προσαρμογής στην Ελλάδα. Δεύτερο, ότι τα αποτελέσματα μέχρι τότε δεν ήταν ικανοποιητικά. Και τρίτο, μου απαριθμούσε η Κομισιόν ε, διάφορα μέτρα τα οποία θα ληφθούν, όπως μονάδες μεγάλων φορολογουμένων, έλεγχος 1.700 ατόμων με μεγάλα περιουσιακά στοιχεία. Αυτά το 2011. Πριν ένα μήνα, κύριε Σεμέτα, δημιούργησε θόρυβο, αρνητικό θόρυβο, στην ελληνική ε, πολιτική ζωή, κοινωνική ζωή, η δήλωση του Υπουργού Οικονομικών της Ελλάδος ότι έναντι της λίστας Φαλσιανή Λαγκάρντ της λίστας των Ελλήνων καταθετών στη Λίχνεστάιν και Λουξεμβούργο της λίστας των Ελλήνων που έχουν μεγάλα κίνητα στο Λονδίνο εν πάση περιπτώσει το μεγάλο πεδίο της φοροδιαφυγής έχουν γίνει ελάχιστα πράγματα αρκεί να σας πω ότι μόνο δύο περιπτώσεις από τις 54.000 της λίστας που έχουν βγάλει χρήματα από την Ελλάδα έχουν ελεγχθεί. Κατόπιν τούτου η ερώτηση είναι απλή. Σε μια περίοδο που οι, ελληνικοί, Έλληνες εργαζόμενοι πληρώνουν νέους φόρους, φορολογούνται ακόμα και οι άνεργοι. Εσείς ως Επίτροπος, ως Επίτροπος αρμόδιος για τα ζητήματα φορολογίας, είστε ικανοποιημένος από την πάταξη της μεγάλης φοροδιαφυγής στην Ελλάδα. Σας ευχαριστώ πολύ. Well, uh, Σας ευχαριστώ πολύ για την ερώτησή σας. Θα γνωρίζετε ότι ε, συνεργαζόμαστε πολύ με τις ε, φορολογικές αρχές της Ελλάδας προκειμένου να μεταρρυθμιστεί ενδελεχώς το σύστημα το φορολογικό στην Ελλάδα και πρέπει να σας πω ότι έχουμε ήδη αρχίσει να βλέπουμε μια σημαντική πρόοδο Συναντήθηκα πρόσφατα με τον Υφυπουργό Οικονομικών, ο οποίος μου παρουσίασε συγκεκριμένα οικονομικά δεδομένα όσον αφορά την εξέλιξη των εσόδων για το κράτος και για πρώτη φορά από την απαρχή της κρίσης βλέπουμε ότι από πλευράς εσόδων, όσον αφορά δηλαδή τον κρατικό προπολογισμό, έχουμε μία πρόοδο πάνω από την τάση που είχε, προ... σημειωθεί στο παρελθόν. Αυτό καταδεικνύει ότι οι προσπάθειες που καταβάλουμε ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τις ελληνικές φορολογικές αρχές αρχίζουν και αποδίδουν κάποιους καρπούς. Τα γνωρίζετε βέβαια πολύ καλά ότι υπάρχουν πολύ διαφορετικοί φορολογικοί κώδικες που έχουν να κάνουν με το προσωπικό εισόδημα, με την προσωπική περιουσία, με την ιδιοκατοίκηση Πολύ διαφορετικοί λοιπόν κώδικες ακόμα πρέπει να μεταρρυθμιστούν και να εγκριθούν. Άλλοι πάλι όμως έχουν ήδη εγκριθεί και θα καταλήξουμε σιγά σιγά σε ένα εντελώ διαφορετικό φορολογικό περιβάλλον στην Ελλάδα. Βλέπω λοιπόν ότι η γενικότερη τάση είναι θετική. Ωστόσο, παραδέχομαι ότι πολλά πράγματα ακόμα πρέπει να γίνουν. Πολλές προσπάθειες ακόμα πρέπει να καταβληθούν και αυτό άλλωστε αναγνωρίζουν και οι ίδιες οι ελληνικές αρχές. Συντοποιούν ότι η εργασία τους αυτή τη στιγμή κινείται στη σωστή κατεύθυνση, αλλά ότι δεν έχει σε καμία περίπτωση ολοκληρωθεί και ότι θα πρέπει να καταβληθούν και επιπρόσθετες προσπάθειες προκειμένου να βελτιωθεί περαιτέρω το τμήμα των εσόδων, των κρατικών αυτών εσόδων. Όσον αφορά τώρα τη λίστα Λαγκάρντ, στην οποία αναφερθήκατε, Προφανώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ένας σημαντικός ισχυρός θεσμός, αλλά είναι τελικά τα κράτη-μέλη αυτά τα οποία πρέπει να καταβάλουν προσπάθειες προκειμένου να χρησιμοποιήσουν τις διαθέσιμες πληροφορίες, τις πληροφορίες που έχουν σε εθνικό επίπεδο. Δεν μπορεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ξεκινήσει μία δικαστική διαδικασία σε ένα εθνικό δικαστήριο όσον αφορά συγκεκριμένες περιπτώσεις όπως αυτή στην οποία αναφερθήκατε ή συγκεκριμένες περιπτώσεις που έχουμε στη λίστα Λαγκάρντ. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι το ζήτημα αυτό αφορά πληροφορίες οι οποίες πρέπει επικοδομητικά να χρησιμοποιηθούν από τις εθνικές αρχές. Πληροφορίες οι οποίες πρέπει να χρησιμοποιήσει η ελληνική κυβέρνηση στα πλαίσια του εθνικού δικαστικού συστήματος. Θα καλούσα λοιπόν τις αρμόδιες εθνικές αρχές να αναλάβουν δράση για το ζήτημα αυτό. Δική τους πάντως είναι η αρμοδιότητα. Αυτή είναι μια σύντομη απάντηση που μπορώ να δώσω στο ερώτημά σας. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Όλοι έχετε αρχίσει από ό,τι κατάλαβα να υποβάλλετε πλέον ερωτήσεις φορολογικής φύσης. Ο Φιλίπ από ό,τι κατάλαβα θέλει να αποχωρήσει, επομένως σας του δώσω αυτή τη στιγμή το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ Κύριε Επίτροπε, θα ήθελα όντω και εγώ να υποβάλω μια ερώτηση φορολογική φύση. Βλέπω ότι οι περισσότεροι πλέον τέτοιε ερωτήσει θέτουν και όχι, τόσο πολλοί ερωτήσει στατιστικού περιεχομένου. Κάποιε σύντομε λοιπόν ερωτήσει θα ήθελα να υποβάλω. Του τελευταίου μήνε γίνανε κάποιε συζητήσει ε, που έχουν να κάνουν με τι συστάσει τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσον αφορά κάποιε μεταρρυθμίσει που πρέπει να γίνουν από τα κράτη-μέλη συστάσεις ε, που γίνονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και έχουν να κάνουν με το υψηλό κόστος εργασίας σε πολλά κράτη-μέλη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λέει ότι θα πρέπει σιγά-σιγά οι φόροι αυτοί να φύγουν από το κόστος εργασίας και να πάνε περισσότερο προς την κατανάλωση. Να υπάρξει αυτό το tax shift, όπως το αποκαλεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πώς όμως θα γίνει αυτό στην πράξη και πώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα υποστηρίξει τα κράτη-μέλη στην προσπάθειά τους αυτή. Η πρώτη μου λοιπόν ερώτηση είναι θα καταφέρει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτίθεται να πει με πιο συγκεκριμένο τρόπο πώς θα βοηθήσει τα κράτη-μέλη να κάνουν αυτό το tax shift. Δεύτερη τώρα ερώτηση. Τους τελευταίους πάλι μήνες, τελευταίες εβδομάδες, ως Ευρωβουλευτής λαμβάνω πάρα πολλές ερωτήσεις που έχουν να κάνουν με τη φορολογία, τη συζήτηση που έχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη φορολογία με τα κράτη-μέλη και τις πολλές δυσκολίε που έχουν εντοπιστεί. Για παράδειγμα, σε πρόσφατη απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου λέγεται ότι ε, η ταξινόμηση των οχημάτων για τα άτομα τα οποία διαβίουν σε δύο διαφορετικές χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να γίνεται σε μία χώρα, πολλοί όμως καλούνται να πληρώσουν δύο φορές τα τέλη ταξινόμηση. Πολλές φορές τα προβλήματα αυτά λύνονται εντελώ διμερεί, σε διμερές επίπεδο με συγχωρείτε. Σε άλλες περιπτώσεις υπάρχουν άνθρωποι, για παράδειγμα που ζουν στο Βέλγιο και στη Γαλλία και οι οποίοι καλούνται να πληρώσουν δύο φορές. Πώς μπορούμε να ευθυγραμμίσουμε περισσότερο την προσέγγιση αυτή σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Υπάρχουν πάρα πολλοί πολίτε οι οποίοι μπερδεύονται όταν βλέπουν ότι σε ορισμένε περιπτώσεις καλούνται να πληρώσουν μία φορά τα τέλη ταξινόμησης, σε άλλε περιπτώσει οφείλουν να τα καταβάλουν δύο φορέ. Ξέρετε ότι έχουμε και τη σχετική απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μπορείτε να αποσαφηνίσετε κάπως τα πράγματα. Τελευταία ερώτηση, μια συζήτηση η οποία γίνεται πάλι στις τελευταίες εβδομάδες, στους τελευταίους μήνες όσον αφορά το φόρο προστιθέμενης αξίας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να αντιμετωπίσουμε την απάτη σχετικά με το ΦΠΑ και ε, όντως δράση έχει, έχετε προσπαθήσει να λάβετε δράση σχετικά τους τελευταίους μήνες. Βλέπουμε όμως ότι υπάρχουν κάποιες εταιρείες οι οποίες βρίσκονται σε δύσκολη θέση γιατί τελικά τα κράτη δεν αποδίδουν, δεν προχωρούν με την επιστροφή του ΦΠΑ προς ορισμένες εταιρείες οι οποίες στη συνέχεια αντιμετωπίζουν πολύ δύσκολα οικονομικά προβλήματα. Μπορείτε να μας ενημερώσετε και επ' αυτού το έχετε ζητήσει το πρόβλημα αυτό, προβλέπονται λύσεις με τα κράτη-μέλη. Σας ευχαριστώ πολύ. Uh, uh, um, ναι. Για το tax shift, η μετακύληση των φόρων από την εργασία στην κατανάλωση. Ε, υπάρχουν πιο συγκεκριμένες συστάσεις. Εξυπακούεται ότι πρέπει να βρούμε μια σωστή ισορροπία ανάμεσα στην εξειδίκευση των συστάσεων που εκδίδουμε και την αρχή της επικουρικότητας που ε, έχει ιδιαίτερο ειδικό βάρος στον τομέα της φορολογίας. Ακόμη και αν πάρουμε τις συστάσεις του περσινού έτους, βλέπουμε ότι έχουμε ε, ε, ειδικές συστάσεις για την εισαγωγή συγκεκριμένων φόρων Βεβαίω έχουμε κατά νου ότι αν εισαχθεί ε, ο εν λόγω φόρο, ε, παραδείγματο χάρη, δεν θα είναι απαραίτητο ε, και δεν θα επιστηρίζει συνολική αύξηση του φορολογικού άχθους, αλλά θα επιτύχει ε, την μετακύληση των φόρων προς ε, τη μετεξέλιξη των φόρων προς φόρους ευνοϊκότερους για την ανάπτυξη. Βεβαίως αυτό επίσης εξυπακούεται Επίσης αυτό σημαίνει μάλλον ε, ότι πρέπει να ξέρουμε προς τα πού θα στραφούμε με την εισαγωγή νέων φόρων. Στην ε, πρόσφατη ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης διαπιστώσαμε ότι αντί να μειωθεί το φορολογικό άχθος επί της εργασίας τα κράτη-μέλη τελικά υιοθέτησαν διαφορετική προσέγγιση, τουλάχιστον κάποια από αυτά, Και γι' αυτό σας είπα ότι στις ειδικέ αναχώρες συστάσεις πρέπει να είμαστε πολύ συγκεκριμένοι για το θέμα της μετεξέλιξης του φορολογικού συστήματος. Για την φορολόγηση τώρα των αυτοκινήτων. Ε, είναι πολύ μακρά η ιστορία που έχουμε σε αυτό το τομέα και αν θυμάμαι καλά το 2005 ήδη κατέθεσε μία πρόταση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να ε, επιληθεί το ζήτημα της ε, διπλής φορολόγησης των αυτοκινήτων. Δυστυχώς όμως ε, τα κράτη-μέλη δεν κατάφεραν να καταλήξουν σε συμφωνία. Ακόμη εξετάζεται το ζήτημα στο Συμβούλιο, αν δεν κάνω λάθος. Εάν το επιθυμούν, τα κράτη-μέλη μπορούν να το επαναφέρουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για να καταλήξουν συμφωνία. Τέσσερα ήταν τα κράτη-μέλη που δεν μπορούσαν να δώσουν το πράσινο φως, αν θυμάμαι καλά. Και γι' αυτό συστήνουμε στα κράτη-μέλη να χρησιμοποιήσουν το πνεύμα της πρότασης της Επιτροπής για να αντεπεξέλθουν στο πρόβλημα της ε, διπλής φορολόγησης θεσπίζοντας εθνικά μέτρα. Κάποια κράτη-μέλη έχουν ένα υψηλό μέρος των εισοδημάτων τους ε, που προέρχονται από τη φυρολόγηση των αυτοκινήτων και ε, δεν ε, είναι ιδιαίτερα πρόθυμα να μεταρρυθμίσουν το φορολογικό του σύστημα. Για τον φόρο προστιθέμενης αξίας και την απόδοσή του. Στην ε, τρέχουσα οικονομική κατάσταση όπου η ταμιακή ροή έχει μεγάλη σημασία για ε, οποιαδήποτε επιχείρηση, μικρή μεγάλη, οι φορολογικές αρχές των κρατών μελών πρέπει να εξασφαλίσουν ότι γίνονται εγκαίρως εμπρόθεσμα οι αποδόσεις, οι επιστροφές ε, ΦΠΑ ξεκινήσαμε μια διαδικασία επί πρόσφατα κατά ενός ε, κράτους μέλους που κατά τη γνώμη μας ε, έχει μια ε, υπερβολικά μακρόχρονη διαδικασία επιστροφής Και ζητήσαμε και από όλα τα κράτη-μέλη να εξετάσουν ε, την διαδικασία τους, ούτως ώστε σε εύλογο χρονικό διάστημα να επιστρέφεται ο φόρος. Ε, κατά τη γνώμη μου αυτό το εύλογο χρονικό διάστημα δεν υπερβαίνει τις 30 ημέρες. Αυτό θα πρέπει να γίνει η τρέχουσα πρακτική, ιδανικά. Πρόεδρος, α, κυκλοφορούν ε, φήμες ότι έχουμε και άλλες ερωτήσεις. για τα στατιστικά δεδομένα. Ε, ο Hans Πίτερ Μάρτιν, ζητώ συγγνώμη που ήρθα τελευταία στιγμή, αλλά ε, στη διακοινοβουλευτική με την Κίνα συγκάλεσαν ε, εκτάκτως μία συνεδρίαση και δυστυχώς δεν μπορώ να παραμείνω. Είμαι σίγουρος ότι θα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση. Επίτροπε, δύο ερωτήσεις. Πρώτον, όσον αφορά την απάτη σχετικά με το φόρο προστιθέμενης αξίας. Μας είπατε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα χάσμα 1,3 δισεκατομμύρια ευρώ. Αν τώρα όλες οι χώρες αποφάσιζαν να φτάσουν στο ποσοστό που έχουμε στη Γερμανία, δηλαδή το 1%, τότε θα είχαμε 15 δισεκατομμύρια επιπλέον 18 εκατομμύρια θα έργα για χώρες όπως η Ιταλία ετήσιο επίπεδο. Θα δούμε τώρα την κατάσταση του χρέους. Αν είναι 150-180 δισεκατομμύρια συν τους στόκους, τότε ούτε η Ιταλία ούτε η Γαλλία θα είχαν κανένα πρόβλημα, εφόσον θα είχαν ένα επιπλέον εισόδημα. Είπατε επίση ότι θα μπορούσαν να βρεθούν και κάποιες λύσεις όσον αφορά τα κρατικά ομόλογα. Συμφωνείτε με την αξιολόγηση που κάνω εγώ ότι δηλαδή η μείωση της απάτης των φόρων προστιθέμενης αξίας θα ήταν ευνοϊκή για την Ευρωπαϊκή Ένωση, για ποιο λόγο όμως οι λύσεις που έχουν προταθεί δεν εφαρμόζονται. Αναφερθήκατε πριν από λίγο σε ένα πρόγραμμα για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης το οποίο αντιστοιχεί περίπου σε 110 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ περίπου είπατε ότι 40 δισεκατομμύρια ευρώ συνδέονται με την καταπολέμηση της απάτης ε, όσον αφορά την πώληση τσιγάρων, όσον αφορά την λαθρεμπορία τσιγάρων. Για ποιο λόγο λοιπόν βλέπουμε τέτοιες μεγάλες ε, αποκλίσεις από το ένα κρατώσει μέλος στο άλλο και για ποιο λόγο τελικά βλέπουμε ότι ορισμένα κράτη-μέλη έχουν ε, πολύ καλύτερες επιδόσεις από ό,τι άλλα. Πώς μπορούμε να γεφυρώσουμε το χάσμα που βλέπουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πώς μπορούμε να ανακτήσουμε το απολεσθέν αυτό εισόδημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το συγκεκριμένο πρόγραμμα στο οποίο αναφερθήκατε, έχει την υποστήριξη και των μεγάλων καπνοβιομηχανιών. Νομίζω λοιπόν ότι θα έπρεπε να λειτουργήσει σωστά εφόσον έχετε μια πολύ στεναρή υποστήριξη. Well, uh, I completely agree. Uh, Συμφωνώ απόλυτα ότι το χάσμα στο φόρο προστιθέμενης αξίας αποτελεί πραγματικά ένα σημαντικότατο πρόβλημα. Και αφού ολοκληρωθεί η όλη ανάλυση και αξιολόγηση, θα πρέπει να πούμε ξεκάθαρα ότι πρέπει να συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας για την καταπολέμηση της απάτης που σχετίζεται με το φόρο προστιθέμενης αξίας. Βρισκόμαστε πάντως στη σωστή κατεύθυνση αυτή τη στιγμή. Αυτός είναι ο στόχος που πρέπει να κυνηγήσουμε. Ωστόσο, από θεωρητικής πλευράς, δεν μπορούμε να πούμε ότι τα 193 δισεκατομμύρια ευρώ συνδέονται αναγκαστικά με την απάτη στο φόρο προστιθέμενης αξίας. Υπάρχουν και κάποιοι άλλοι παράγοντες που πρέπει να ληφθούν υπόψη, όπως η χροκοπία ορισμένων εταιριών ή οι καθυστερήσεις στην καταβολή του φόρου προστιθέμενης αξίας ορισμένες περιπτώσεις. Οι συνιστώσεις αυτές συμβάλλουν στο σημαντικότατο αυτό ποσό, αλλά θα έλεγα ότι το σημαντικότατο μερίδιο οφείλεται στην απάτη σχετικά με το φόρο προστιθέμενης αξίας. Ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήδη έχουμε παρουσιάσει τα μέτρα τα οποία μπορούμε να εφαρμόσουμε στο στάδιο αυτό και χάρη στην πολύ ταχύ εργασία που έγινε στον τομέα αυτό καταλήξαμε συμφωνία με τα κράτη-μέλη για ένα μηχανισμό έγκαιρη ε, ανάληψης δράσης για την αντιμετώπιση τη απάτης στο φόρο προστιθέμενης αξίας. Είπαμε επίσης ότι θα πρέπει να υπάρχει μια επέκταση του μηχανισμού αντιστροφής του βάρου προκειμένου να καταφέρουμε να προωθήσουμε περισσότερο την πρόθεση των προϊόντων και των υπηρεσιών. Να μην επιβαρύνεται δηλαδή αυτό ο τομέα. Και υπάρχουν όντω κάποια κράτη-μέλη τα οποία ήδη έχουν αρχίσει να χρησιμοποιούν το μέσο αυτό για να αντιμετωπίσουν τη διασυνοριακή επάτη στο φόρο προστιθέμενη αξία. Παράλληλα, συνεχίζουμε την εργασία μα προκειμένου να καταλήξουμε σε ένα οριστικό καθεστώ φόρου προστιθέμενη αξία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό άλλωστε υποσχεθήκαμε στη γενικότερη στρατηγική μα για το φόρο προστιθέμενη αξία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και, κατά την άποψή μου, όταν καταφέρουμε τελικά να πετύχουμε μια οριστική συμφωνία για ένα ενιαίο καθεστώ φόρου προσθεμένη αξία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τότε και μόνο τότε θα μα εφέσει να αντιμετωπίσουμε τα περισσότερα προβλήματα τα οποία έχουν να κάνουν με τη διασυνοριακή απάτη στο φόρο προσθεμένη αξία. Παράλληλα, βλέπουμε ότι η απάτη αυτή δεν συνδέεται μόνο με τις διασυνοριακές συναλλαγές, αλλά και σε εθνικό εσωτερικό επίπεδο λαμβάνει η χώρα η απάτη αυτή, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι τα κράτη-μέλη οφείλουν και τα ίδια να υιοθετήσουν εθνικά μέτρα για να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα αυτό. Πρόσφατα μάλιστα <coughs> είχαμε μια πολύ επικοδομητική συνδιάσκεψη ειδικά για τα προβλήματα συλλογής φόρου προστιθέμενης αξίας, όπου ορισμένα κράτη-μέλη παρουσίασαν ιδιαίτερα καινοτόμες θα έλεγα πολιτικές για την βελτίωση της, του συστήματος συλλογής φόρου προστιθέμενης αξίας. Η Πορτογαλία, για παράδειγμα, έχει εισάγει ένα εντελώς νέο σύστημα για τη συλλογή του φόρου προστιθέμενης αξίας, χρησιμοποιώντας ένα μοντέλο το οποίο εμεί προτείναμε ω Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην πράσινη βίβλο μα πριν από μερικά χρόνια. Έχουν αρχίσει λοιπόν οι Πορτογάλοι να το εφαρμόζουν αυτό στην πράξη και έκτοτε έχουν δει ότι έχουν αυξηθεί πάρα πολύ τα κρατικά έσοδα τα οποία απορρέουν από τη συλλογή του φόρου προσεθεμένης αξίας. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι μπορούν τα ίδια τα κράτη-μέλη να εμπνευστούν από τις βέλτιστες πρακτικές που υπάρχουν σε άλλα κράτη-μέλη και να εφαρμόσουν και αυτά σε εσωτερικό επίπεδο τέτοια μέτρα. Τώρα, όσον αφορά το ζήτημα της προστασίας των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επ' αυτού θα ήθελα πάλι να είμαι ιδιαίτερα σαφής. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε να συμπεριλάβει το φόρο προστιθέμενης αξίας ως τομέα αρμοδιότητας του κανονισμού αυτού για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το σχετικό δίκαιο που θα πρέπει να διέπει, ποινικό δίκαιο που θα πρέπει να διέπει τον κανονισμό αυτό. Δυστυχώς πολλά κράτη-μέλη αποφάσισαν να αποκλείσουν το φόρο προστιθέμενης αξίας. Επομένως αποκλείεται από την οδηγία, από την οδηγία αυτή. Θα ήθελα λοιπόν να ζητήσω από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να τοποθετηθεί στεναρά και όταν θα διαπραγματευόμαστε την οδηγία αυτή καθ' αυτή θα ήθελα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να ζητήσει να συμπεριληφθεί εκ νέου ο τομέας του φόρου προστιθέμενης αξίας σε αυτή την οδηγία. Κατά αυτόν τον τρόπο θα έχουμε τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουμε ποινικέ διαδικασίες για την καταπολέμηση της απάτης του φόρου προστιθέμενης αξίας. Ολοκληρώνοντας, θα ήθελα να σας πω ότι η εργασία που κάνουμε αυτή τη στιγμή με τα κράτη-μέλη βρίσκεται στο σωστό δρόμο και θα πρέπει να ξέρετε ότι στον τομέα της φορολογίας όπως και στον τομέα του φόρου της αξίας ισχύου κανόνας της ομοφωνίας και ως εκ τούτου ακόμα και αν καταβάλουμε εμείς πολύ σημαντικές προσπάθειες η τελική απόφαση εξαρτάται από τα κράτη-μέλη. Θα ήθελα λοιπόν να ζητήσω από τα κράτη-μέλη να υποστηρίξουν περισσότερο τις πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε αυτό το συγκεκριμένο τομέα. Uh, Ευχαριστώ. Βέρνε, είσαι ο επόμενος. Μου έχεις και εσύ καμία μια φορολογική ερώτηση. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κοιτάξτε, επειδή βλέπω τώρα πως ε, έχουμε ένα ζήτημα το οποίο από ό,τι φαίνεται θα μας απασχολήσει ενώπιση των εκλογών. Κοιτάξτε, έχετε κάνει μια πρόταση από πλευράς Κομισιόν να ενισχυθούν οι ε, αρμοδιότητες Κομισιόν. Έχουμε εθνικούς ε, εγωισμούς και από τη χώρα μου, λανθασμένες πληροφορίες όχι μόνο από την Ελλάδα και από άλλες χώρες. Τώρα ενισχύσαμε την Eurostat ε, και το ερώτημά μου είναι ποια προβλήματα εξακολουθούν να υπάρχουν με τα κράτη-μέλη. Ε, είναι επαρκής η συνεργασία σας. Θέλουν ε, εγκαίρως τα στοιχεία. Ποιες δυνατότητες κυρώσεις, κυρώσεων έχετε. Και τελικά ποιος ε, είναι αρμόδιος για τα στοιχεία αυτά της Eurostat. Είναι και τα κρατημέλη ή μόνο η Κομισιόν. Μάλιστα, ε, επιτέλους μια ερώτηση για τη στατιστική. Κοιτάξτε. Έπνεμε σαφής ε, με την έγκριση της ε, νομοθεσίας για τα ηλεκτρονικά στατιστικά στοιχεία η κατάσταση έχει βελτιωθεί δραματικά. Και Για την εφαρμογή της νέας νομοθεσίας ε, ενισχύσαμε και τις δυνατότητες της Eurostat από πλευράς ανθρωπίνων πόρων ε, και τώρα έχουμε πολύ περισσότερους ανθρώπους που ασχολούνται με αυτό το ζήτημα και μέχρι στιγμής θεωρώ πως ε, η δουλειά που γίνεται με τα κράτη-μέλη με επαλήθευση των δεδομένων όταν αυτό χρειάζεται μας επιτρέπει να διασφαλίσουμε πως έχουμε στατιστικά στοιχεία υψηλής ποιότητας και αν δείτε την ε, τελευταία Ε, τα τελευταία δελτία στατιστικών στοιχείων ε, έχουμε μόνο μία επιφύλαξη από πλευράς Eurostat. Αν θυμάμαι καλά αφορούσε την Αυστρία λόγω ενός συγκεκριμένου ζητήματος ε, σε επίπεδο κάτω του εθνικού. Ένα θέμα το οποίο νομίζω αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή και η Εθνική Στατιστική Αρχή και η Eurostat. Αυτό αποδεικνύει νομίζω πως η σχετική νομοθεσία λειτουργεί. Υπάρχει ένα άλλο τμήμα των στατιστικών στοιχείων που είναι επίσης σημαντικό από την Ευρωπαϊκή Σκοπιά και αφορά τις μακροοικονομικές ανισορροπίες και τη διαδικασία. Τη σχετική για μένα είναι εξαιρετικά σημαντικό. Εγώ θεωρώ πως εάν είχαμε, είχαμε αυτή τη διαδικασία πριν από 10 χρόνια, πιθανώς αυτή η κρίση να μην ήταν τόσο βαθιά όσο είναι. Και βεβαίως ε, είναι σημαντικό το ότι η διαδικασία αυτή βασίζεται σε στατιστικά δεδομένα υψηλής ποιότητας και εκεί πέρα οι αρμοδιότητες της Eurostat αυτή τη στιγμή είναι πολύ πιο περιορισμένες ε, από ότι στον τομέα των ε, στατιστικών στοιχείων. Γι' αυτό κάναμε πρόταση ακριβώς για τον κανονισμό των ε, ανισορροπιών αυτών για να υπάρχει ακριβώς να υπάρχουν ίδιες αρμοδιότητες μεταξύ των οποίων και οι κυρώσεις που θα μπορούσαν να ισχύσουν που ισχύουν με στην περίπτωση των ε, στατιστικών στοιχείων αλλά όχι στην περίπτωση των ανισορροπιών, των ανισορροπιών όπως είπαμε. Σε περίπτωση κάποιο κράτος μέλος ε, χειραγωγεί τα δεδομένα όπως ξέρετε υπάρχει αυτή η δυνατότητα οπότε Ελπίζω λοιπόν να υιοθετηθεί ο φιλόδοξος σχετικός κανονισμός και έτσι από πλευράς οικονομικής διακυβέρνησης Ευρωπαϊκής Ένωσης θα έχουμε νομίζω στατιστικά δεδομένα υψηλής ποιότητας και επαρκή μέσα στα χέρια της Eurostat για να αντιμετωπίσουμε ζητήματα στα κρατημέλη αν αυτά προκύψουν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να συγχωρείτε για το πώς είχε η σειρά των ερωτήσεων μας ε, και το ότι δεν αφορούσαν το θέμα. Βεβαίως μας ενδιαφέρει η ακρίβεια των στατιστικών στοιχείων και Οπότε φαίνεται θα θυμάστε πως είχαμε Είχατε και στις 8 με 10 προτάσεις κάνει σχετικά με τα σατσικαστία και είστε πολύ δραστηροί, το εκτιμούμε. <coughs> Υπάρχουν τόσες πολλές ερωτήσεις, ε, ίσως γιατί από ό,τι φαίνεται δουλεύει το σύστημα. Τώρα περνάμε στην φορολογία. Μπορείτε λοιπόν να απαντήσετε και σε αυτές τις ερωτήσεις, θα έχουμε φαντάζομαι και άλλες. Δεν ξέρω, ίσως να θέλετε να προσθέσετε κάποια πράγματα και για, τα, για τη στατιστική. Και με συγχωρείτε που έλειπα από την παρουσίασή σας. Λοιπόν, κύριε Επίτροπε, σας ευχαριστώ, Σάρον. Αν συμφωνείτε θα κάνω μια σύντομη εισαγωγή και μετά θα απαντήσω στις ερωτήσεις. Είχα έρθει εδώ πέρα τελευταία φορά τον Μάιο όταν ανέπτυξα τις ιδέες μου για ε, εντονότερη καταπολέμηση της φορολογικής απάτης και της ε, φοροδιαφυγής. Στο διεθνές επίπεδο, με τη στήριξη των G8 και G20, έχει γίνει δεκτή η αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών παγκοσμίω και το σχέδιο δράσης του ΟΣΑ, το λεγόμενο BEPS, για την μείωση της φορολογικής ε, βάσης, έχει εγκριθεί ως μια διεθνής απάντηση στον επιθετικό φορολογικό σχεδιασμό και την εταιρική φοροδιαφυγή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έπαιξε ένα κέριο ρόλο στο να δεσμευτούν οι ηγέτες του κόσμου για να βελτιωθεί η παγκόσμια φορολογική διοίκηση. Για μένα αυτό είναι απόδειξη ότι μπορεί να επιτευχθεί όταν εργαζόμαστε ως Ένωση. Αλλά δεν έχουμε ακόμα τελειώσει. Αύριο πάω στην Αυστραλία, την επόμενη χώρα η οποία θα έχει την προεδρία των G20 και θα μεταφέρω τις προσδοκίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μια ισχυρή πολιτική κατεύθυνση από πλευράς τους για να μην μειωθεί η πίεση κατά της διεθνούς φοροδιαφυγής. Εν μεταξύ, στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επίσης είχαμε ένα παραγωγικό εξάμεινο. Οι νέες πρωτοβουλίες ε, που έχουν αληθεί είναι εντυπωσιακέ. Από το Μάιο είχαμε πρόταση επέκτασης της αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών εντός Ένωσης, συμφωνία σε ένα μηχανισμό γρήγορη αντίδραση καταπολέμησης απάτη του ΦΠΑ. Ξεκινήσαμε διαπραγματεύσει για ισχυρότερε φορολογικέ φωνίε με του γείτονέ μα. Ξεκίνησε η συζήτηση φορολογία τη ψηφιακή οικονομία. Ε, Επίση, ε, προτάθηκε ένα ενιαίο έντυπο ΦΠΑ για να βελτιωθεί η συμμόρφωση και μόλις χτες προτείναμε τροποποιήσεις στην οδηγία μητρικής θηγατρικής για να μην υπάρχει κατάχρηση του φορολογικού συστήματος. Η Κομισιόν έχει χρησιμοποιήσει κάθε εργαλείο στη διάθεσή της για να προωθήσει τις αρχές της ορθής διοίκησης. Εν τω μεταξύ, οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στήριξαν πλήρως ε, τις ε, φιλοδοξίες μας αυτές στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Μαΐου και απέτησαν σαφή πρόοδο και αποτελέσματα. Οπωσδήποτε θα γνωρίζετε πως ακόμη μια φορά το Συμβούλιο ΕΚΟΦΗΝ δεν κατέληξε συμφωνία για την οδηγία αποταμιεύσεων. Αναλήφθηκε το Μάιο μία δέσμευση να συμφωνήσουμε επί του θέματος αυτού μέχρι το τέλος του έτους και πρέπει να την τηρήσουμε. Θα επαναλάβω στους Υπουργούς Οικονομικών τον Δεκέμβριο πως ο κόσμος προχωράει στην αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών και δεν πρέπει να μείνουμε πίσω. Θα ήθελα επίσης να σας ενημερώσω πως οι διαπραγματεύσεις με το Μονακό, την Ανδόρα, το Λιχτενστάιν και το Σαν Μαρίνο έχουν ήδη ξεκινήσει και προχωρούν ικανοποιητικά. Και θα ξεκινήσουμε με την Ελβετία μόλις έχουν και αυτή την δική τους διαπραγματευτική εντολή τις επόμενες εβδομάδες. Τώρα, στην σχετική αλλά χωριστή πρόταση για την οδηγία διοικητική συνεργασίας. Ελπίζω το Κοινοβούλιο να στηρίξει πλήρως ε, το διευρυμένο πεδίο εφαρμογής περί ανταλλαγής πληροφοριών όταν θα ψηφιστεί στην Ολομέλεια του Δεκεμβρίου το θέμα αυτό. Επίσης, η καταπολέμηση της φοροδιαφυγής ανέδειξε νέες και ενδιαφέρουσες προκλήσεις. Μεταξύ αυτών το πώς θα φορολογηθεί η ψηφιακή οικονομία με τρόπο δίκαιο χωρίς να εμποδιστεί η ανάπτυξη του σημαντικού αυτού κλάδου. Αλλά το ότι ο κλάδος αυτός είναι νέος και τα μοναδικά του χαρακτηριστικά σημαίνει πως δεν υπάρχει κάποια εμπειρία στην οποία μπορούμε να βασιστούμε όσον αφορά την φορολογία του. Δεν υπάρχουν εύκολες απαντήσεις ή γρήγορες λύσεις. Γι' αυτό συστήσαμε μία ομάδα ειδικών υψηλού επίπεδου για να βρουν τις βασικές προκλήσεις που σχετίζονται με την ε, ψηφιακή ε, φορολογία και να παρουσιάσουν λύσεις μέχρι το καλοκαίρι του επόμενου έτους. Η τελική επιλογή των μελών της ομάδας αυτής ε, με μέλη από και τον φορολογικό κλάδο και τον ψηφιακό κλάδο ανακοινώθηκε χτες. Πρόεδρος θα είναι ο Βίκτορ Γκάσπαρ, πρώην Πορτογάλος Υπουργός Οικονομικών, ο οποίος απολαμβάνει τις πληρούς εμπιστοσύνη μου. Ένα άλλο θέμα μεγάλης σημασίας είναι η καταπολέμηση της φοροδιαφυγής ε, στον τομέα του ΦΠΑ. Θα ήθελα επί να ευχαριστήσω την Σάρον Μπόουλς για τη συμμετοχή της στο φορολογικό φόρουμ των Βρυξελών την προηγούμενη εβδομάδα όπου συζητήθηκε ο ΦΠΑ. Στόχος μας είναι ένα πιο αποτελεσματικό και εύρωστο σύστημα ΦΠΑ. Τον Οκτώβριο η Κομισιόν δημοσίευσε μια έκθεση για το χάσμα του ΦΠΑ στην Ευρώπη, το οποίο υπολογίζεται σε 193 δισεκατομμύρια ευρώ το 2011. ένα ανησυχητικό νούμερο, το οποίο επίσης επιβεβαιώνει πως η μεταρρύθμισή μας πηγαίνει προς σωστή κατεύθυνση. Το να κλείσουμε αυτό το χάσμα του ΦΠΑ σημαίνει εντατικοποίηση και της καταπολέμησης της απάτης και βεβαίως να διευκολύνουμε όσους θέλουν να συμμορφωθούν αλλά αντιμετωπίζουν την πολυπλοκότητα του συστήματος. Και στα δύο αυτά μέτωπα έχουμε επιτύχει πρόοδο σημαντικά νέα μέτρα έχουν ληφθεί για να καταπολεμηθεί η απάτη του ΦΠΑ, κυρίως με την υιοθέτηση του μηχανισμού γρήγορης αντίδρασης. Επίσης, σημαντικά βήματα έχουν αναλυφθεί για να μειωθεί η γραφειοκρατία για επιχειρήσεις και να διευκολυνθεί η συμμόρφωση. Η τυποποιημένη δήλωση ΦΠΑ θα μειώσει το κόστος για τις επιχειρήσεις κατά 15 δισεκατομμύρια ευρώ το έτος και θα διευκολύνει την υποβολή δηλώσεων ΦΠΑ σε ολόκληρη την Ένωση. Θα ήθελα να ευχαριστήσω εδώ πέρα τον κύριο Στρέιτσεκ για την έκθεσή του. Η αναθεώρηση του γενικού συστήματος του ποσοστού ΦΠΑ αυτή τη στιγμή είναι εν εξελίξη. Είχαμε πάρα πολλέ συνεισφορέ από ενδιαφερόμενου και ειδικού. Δεν έχουμε ακόμη βγάλει κάποια συμπεράσματα. Το επόμενο βήμα θα είναι μια αξιολόγηση αντικτύπου αρχέ του επόμενου έτου που θα μας βοηθήσει να βρούμε την σωστή ε, προσέγγιση. Τώρα θα ήθελα να αφαιρθώ σε κάποια άλλα ζητήματα στα οποία θα ήθελα να έχουμε κάποια πρόοδο. Ξεκινώντας με την ε, κοινή φορολογική βάση. Προχωράμε σε τεχνικό επίπεδο, αλλά για να είμαι ειλικρινής, δεν είναι ικανοποιητικός ο ρυθμός των συζητήσεων. Πρέπει να περάσουμε σε μια πραγματική πολιτική συζήτηση για την κοινή εταιρική φορολογική βάση, δεδομένης της σημασίας της ε, στο ε, ευρύτερο πλαίσιο της ε, εταιρικής φοροδιαφυγής. Οπότε πρέπει να υπάρξει κάποια πολιτική όθηση, αν είναι να μην χάσουμε το τρένο. Τώρα, στον φόρο χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, Τώρα πρέπει τα 11 κράτη-μέλη να κινηθούν γρήγορα. Δεν θα κερδίσουμε τίποτα με τις καθυστερήσεις. Η Κομισιόν έκανε ό,τι μπορούσε για να υποστηρίξει τις διαπραγματεύσεις και ήταν ιδιαίτερα επικοδομητική και η στάση του Κοινοβουλίου. Πάρα πολλέ λογικές λύσεις ε, είναι προς συζήτηση. Τώρα πρέπει να υπάρξει μια πολιτική όθηση. Τέλος, για την ε, οδηγία φορολόγησης ενέργειας φοβάμαι πως χάνουμε εδώ πέρα μια σημαντική ευκαιρία. Τα τελευταία συμβαστικά κείμενα είναι δυστυχώ καθόλου φιλόδοξα. Η Κομισιόν αυτή τη στιγμή αναζητά λύσει για το θέμα αυτό. Κυρίε και κύριοι βουλευτές, όπως ξέρετε, ο κατάλογος των νέων προτάσεων του 2014 είναι πάρα πολύ μικρός, καθώς η θητεία και της Κομισιόν και του Κοινοβουλίου λίγη. Αυτό όμω δεν σημαίνει πω σταματάει η δουλειά μα, αντιθέτω έχουμε πάρα πολλά πράγματα πρέπει να γίνουν τους επόμενους 12 μήνες. Γι' αυτό πρέπει να προωθήσουμε όλα τα ανοιχτά μέτωπα, να διατηρηθεί η ορμή όπου αυτή υπάρχει και να δώσουμε όθηση εκεί όπου δεν υπάρχει. Παραδείγματο χάρη τα εργαλεία για καλύτερη καταπολέμηση της φοροδιαφυγής υπάρχουν και η πολιτική βούληση. Τώρα πρέπει τα κράτη-μέλη να διατηρήσουν το ρυθμό που υπάρχει και να καταλήξουν στα συγκεκριμένα μέτρα τα οποία χρειάζονται. Όσον αφορά το ΦΠΑ, πρέπει να γίνει περισσότερη δουλειά. Κατά διάρκεια του επόμενου έτους πρέπει να βρεθεί μια λευκή βίβλος η οποία θα υιοθετηθεί για ένα οριστικό καστό ΦΠΑ για τις ε, διασυνοριακές ε, προμήθειες αγαθών. Θα ήθελα λοιπόν να ακούσω τις δικές σας απόψεις για το πώς βλέπετε να προχωρούν τα πράγματα και το τι περιμένετε. Σας ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Δεν έχει ζητήσει κάποιος... Δεν έχει έρθει κάποιος ακόμα από το ΕΛΚ. Αστρίντ, είστε έτοιμοι να κάνετε ερώτηση. Όχι. Η Μαριάν πρώτη. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, ευχαριστώ που ήρθατε και μας ενημερώσατε. Αλλά δεν μπορούμε να μιλάμε για συγκεκριμένα αποτελέσματα σε όλα τα μέτωπα. Σας ευχαριστώ για τις προσπάθειες που έχετε κάνει. Αλλά η φορολογική απάτη είναι ένα θέμα πάρα πολύ ευαίσθητο. Κανείς δεν θέλει διπλή φορολογία, αλλά δεν θέλει και να ξεφεύγουν κάποιοι. Για την πρόταση που κάνατε χτες για την ε, μητρική και θυγατρική εταιρεία, και εδώ πέρα, ναι εντάξει να αποφύγουμε τη διπλή φορολογία, αλλά πρέπει να μην υπάρχει και φοροαποφυγή μέσω διαφόρων ε, συναλλαγών εντός του ιδίου ομίλου. Και αυτό δεν είναι αποδεκτό. Πρέπει λοιπόν να γίνει κάτι αποτελεσματικό. Δεν έχουμε δει ακόμα την πρόταση, αλλά επί της αρχής ε, την στηρίζουμε. Αλλά να σας ρωτήσω το εξής. Ε, τι γίνεται στο ΕΚΟΦΗΝ, τι στάση έχουν τα κράτη-μέλη, γιατί και εδώ πέρα χρειάζεται συνένεση, έτσι. Όταν λέτε πως πρέπει να έχει τελειώσει τέλος του 2014, είναι ρεαλιστικό, το πιστεύετε ότι θα γίνει. Γιατί ε, το βλέπουμε, όπως και με τις τράπεζες, όπως και με άλλα μεγάλα πακέτα, ο κόσμος θέλει να κάνουμε κάτι, ε, λέμε πως ε, δουλεύουμε πάνω στο θέμα, αλλά δεν βλέπουν αποτελέσματα. Και ξέρω πως ε, βεβαίως ε, αυτά τα πράγματα δεν γίνονται από τη μια μέρα στην άλλη. Έχετε ενέργεια, ελπίζω λοιπόν πριν από τις εκλογές να έχουμε κάποια συγκεκριμένα αποτελέσματα τα οποία θα είναι απτά. Δεύτερο ερώτημα το οποίο αφορά ακριβώς την κοινή εταιρική φορολογική βάση. Είχαμε κάνει μια έκθεση εδώ πέρα στο Κοινοβούλιο και έχουμε ένα συγκεκριμένο ε, χρήσιμο εργαλείο για τις επιχειρήσεις που σημαίνει πράγματι απλούστευση του διοικητικού βάρους αλλά έχουμε ένα μέσο το οποίο επίσης θα καταπολεμήσει την φοροαποφυγή και θα επιτρέψει να φορολογούνται επιχειρήσεις εκεί όπου κανονικά θα έπρεπε να φορολογούνται. Πώς έχουν λοιπόν τα πράγματα με το θέμα αυτό οι επαφές μου με ανθρώπους που είναι στις ομάδες εργασίας μου λένε πως έχουν μπει στην τεχνική και δύσκολη δουλειά γιατί βεβαίως δεν είναι καθόλου απλή αυτή η υπόθεση αλλά θεωρείτε πως θα έχουμε κάποια πολιτική απόφαση εντός αυτής της ε, θητείας ή δεν θα τα καταφέρουμε. Ευχαριστώ. Thank Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω τη Μαρία Τάισεν. Είναι εξαιρετική η έκθεσή σας για το CCTV. Όπως είπα και στην εισαγωγική μου παρουσίαση, θα ήθελα να επιταχυνθεί η πρόοδος που σημειώνεται σε αυτό το τομέα. Νομίζω δίκιο είχατε όταν στην έκθεσή σας αναφέρατε πως πρέπει να είναι δεσμευτική διάταξη για τις πολυεθνικές εταιρείες από ένα όριο και πάνω. πέρα από την μείωση του άχθους που ήταν ο αρχικός στόχος της πρότασης. Υπάρχουν και άλλα ζητήματα που σχετίζονται με τη φορά απόφυγη και διαφυγή. Κατά τη γνώμη μου θα ήταν ε, εποφελής ε, η λύση αυτή και για τις δύο πλευρές. Και γι' αυτό ε, συνεχίζω να σκοπίεση. συζήτησα με τις επερχόμενες προεδρίες, την ελληνική και την ιταλική, και χαίρομαι που κρίνουν ότι είναι ε, προτεραιότητα ο φάκελος αυτός και για τις δύο προεδρίες. και ε, ε, ευελπιστώ ότι από το τεχνικό πεδίο θα μπορέσουμε να σπρώξουμε αυτήν τη συζήτηση στο ΕΚΟΦΗΝ και άρα σε πιο πολιτικό επίπεδο. Κατά πάσα πιθανότητα θα γίνει αυτό στην ε, Προεδρία. Φυσικά αυτό θα εξαρτηθεί και από την πολιτική καθοδήγηση που θα δοθεί ε, από το ΕΚΟΦΗΝ και θα συνεχιστούν οι εργασίες στην Ιταλική Προεδρία. Πάντως η εταιρική φορολόγηση, δίκιο έχετε, είναι ένα εξαιρετικά περίπλοκο δύσκολο ζήτημα και ε, υπάρχει μια πληθώρα τεχνικών ζητημάτων που πρέπει να αξιολογηθούν και να αναλυθούν επακριβώς και να γίνουν αντιληπτά με τον ίδιο τρόπο από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Αυτό είναι χρονοβόρο. Πάντως, ε, στο πολιτικό θεματολόγιο του ΕΚΟΦΗΝ ελπίζουμε να προσθεθεί αυτό το ζήτημα και ξαναλέω ελπίζουμε να γίνει αυτό στην Ελληνική Προεδρία. Σε σχέση με τις διασυνοριακές ε, δραστηριότητες των ε, μητρικών και θηγατρικών ε, εταιριών, εχθές Κάναμε μια πρόταση οδηγίας για τις μητρικές θηγατρικές που έχει ιδιαίτερη σημασία διότι εξετάζει αυτά τα συγκεκριμένα διασυνοριακά ζητήματα μητρικών που έχουν πολλαπλές θηγατρικές και τα δύο ε, στοιχεία έχουν ιδιαίτερη σημασία. Τα υβριδικά δάνεια είναι κατά τη δική μας αξιολόγηση είναι ένα ευρέως διαδεδομένο φαινόμενο και χρησιμοποιούνται για λόγους φοροαποφυγής από τις πολυεθνικές. Θα κλείσουμε αυτό το παραθυράκι αν εγκριθεί η οδηγία από τα κράτη-μέλη. Πέραν αυτού υπάρχει και ο κανόνας ε, κατά της καταχρηστικής συμπεριφοράς. Προτείνεται και αυτό μέσα στην οδηγία. Μας επιτρέπει να αντιμετωπίζουμε καταστάσεις όπου η ενιαία μας αγορά ε, επηρεάζεται από τις διμερείς σχέσεις των κρατών μελών με τρίτες χώρες. Φυσικά, το θέμα τίθεται όταν σε συνδυασμό με τις διμερείς ε, συμφωνίες των κρατών μελών της Ένωσης ε, για διπλή φορολόγηση ε, δημιουργούν προβλήματα επίσης φορολόγησης στην Ένωση ως ενιαία αγορά. Οπότε η καταπολέμηση αυτής της καταχρηστικής συμπεριφοράς μέσω των διατάξεων της οδηγίας θα μας επιτρέψει να θέσουμε υποέλεγχο έλεγχο αυτές τις συναλλαγές. Ε, σε περίπτωση που δημιουργείται μια δομή ε, ακριβώς για να ε, διοχετευθούν τα κέρδη σε φορολογικές επικράτειες όπου δεν είναι εφαρμοστές οι ίδιες φορολογικές διατάξεις και δεν είναι φορολογητέα ύλη τα κέρδη. Στο ΕΚΟΦΗΝ νομίζω ξεκάθαρα φάνηκε ότι οι Υπουργοί Οικονομικών έχουν αναλάβει ισχυρή δέσμευση για να αντιμετωπίσουν το θέμα της ποροδιαφυγής φοροδιαφυγής. Και συζητήσεις που είχα με τους Υπουργούς ξεκάθαρα είπανε ήρθε η στιγμή να ε, έχουμε αποτελέσματα. Δεν αρκεί πλέον να λέμε ότι θέλουμε να αντιμετωπιστεί το ζήτημα. Έχουμε όλα τα χρειαζόμενα στη διάθεσή μας. Ε, και αυτό που χρειαζόμαστε είναι να εγκριθούν οι προτάσεις που έχουν γίνει και στην πράξη να αποδείξουμε ότι δεν παραμένουμε στα λόγια αλλά περνάμε και στα έργα είναι πια το, θέμα στα χέρια των Υπουργών στο ΕΚΟΦΗΝ. Ελπίζω να κάνουν τα, αυτά που πρέπει. σε ευχαριστώ. Για τους σοσιαλιστές η κυρία Κλέβερ. Ευχαριστώ. Κύριε Επίτροπε, καλώς ήρθατε πάλι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στην Επιτροπή μας. Συμφωνώ μαζί σας ότι δεν θα πρέπει να σταματήσουμε τον αγώνα κατά των φοροφυγάδων και της φοροδιαφυγής. Θα πρέπει να αναλάβουμε πιο ενεργό ρόλο και να θέσουμε ως προτεραιότητα στην πολιτική ατζέντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης το ζήτημα αυτό. Γι' αυτό το λόγο στην Ολομέλεια του Κοινοβουλίου το Δεκέμβριο θα υπάρχει ένα κοινό ψήφισμα όσον αφορά τις μετρήσιμες και δεσμευτικές, τα δεσμευτικά μέτρα για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής. Γνωρίζουμε ότι υπάρχει ένα σχέδιο δράσης Ευρωπαϊκής Επιτροπής εδώ και ένα χρόνο και ότι γίνονται και δύο συστάσεις όσον αφορά την, τον επιθετικό φορολογικό σχεδιασμό καθώς επίσης και τους φορολογικούς παραδείσους. Δυστυχώς όμως δεν είδαμε τα αναμενόμενα αποτελέσματα και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εγκρίναμε και το Μάιο μία έκθεση για τα ζητήματα αυτά. Εγκρίθηκε συγκεκριμένα το Μάιο. Πολύ καλό το κείμενο αυτό αλλά και πάλι δεν ήταν δεσμευτικό. Καταφέραμε ωστόσο στο Συμβούλιο να επηρεάσουμε τα πράγματα προς το δικό μας μέρος, προς τη δική μας την κατεύθυνση. Αλλά και πάλι δεν έχουν γίνει πάρα πολλά πράγματα όσον αφορά την νομοθετική δράση που πρέπει να λάβει η χώρα για συγκεκριμένες πλέον δεσμεύσεις, για δεσμευτικές διατάξεις. Θέλουμε να υπάρχουν πραγματικές δεσμεύσεις από τα κράτη-μέλη προκειμένου να μειωθεί το φορολογικό χάσμα. Στα κράτη-μέλη που ανέλαβαν τέτοια δράση έχουμε δει σημαντική πρόοδο όσον αφορά την πάταξη της φοροδιαφυγής. Η ερώτησή μου είναι η ακόλουθη. Κύριε Επίτροπε, μπορούμε να έχουμε σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο μια ομάδα δικτών που θα βοηθούσαν τα κράτη-μέλη να επικεντρωθούν περισσότερο στην γεφύρωση του φορολογικού χάσματος και ποια συγκεκριμένα μέτρα μπορείτε εσεί να αναλάβετε προκειμένου να γεφυρωθεί το φορολογικό αυτοχάσμα ιδίω στα πλαίσια του ευρωπαϊκού εξαμήνου και στα πλαίσια της στρατηγικής Ευρώπη 2020 που ε, εν τέλει είναι η βασική ε, στρατηγική καθοδήγηση στην οποία έχουμε. Καταρχάς, να ευχαριστήσω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την στεναρή υποστήριξή του σε όλες τις δικές μας ε, ενέργειες για το ότι πολλές φορές έχει αναλάβει μια προληπτική δράση για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής αυτό καταλαβαίνετε ότι μας βοηθάει πάρα πολύ να διατηρήσουμε την δυναμικότητα, το δυναμικό χαρακτήρα της όλης αυτής προσπάθειας και μας επιτρέπει να συνεχίζουμε να αναλαμβάνουμε δράση για την πάταξη των φαινομένων αυτών. Όπως είπατε κι εσείς, απομένουν ακόμα πολλά πράγματα τα οποία πρέπει να εφαρμοστούν. Εγώ πιστεύω ότι έχουμε πλέον όλα τα απαραίτητα στοιχεία επιτάπητος και επομένως αν τα κράτη-μέλη εγκρίνουν τα όσα έχουμε προτείνει εμείς, τότε θα σημειωθεί τεράστια πρόοδος στον τομέα αυτό. Και αυτό είναι άλλωστε και προς το συμφέρον των ίδιων των κρατών μελών. Δηλαδή, αν εφαρμοστούν τα μέτρα αυτά, αν εγκριθούν και εφαρμοστούν, θα καταφέρουν να συλλέγουν καλύτερα τους φόρους. Πολλά από αυτά τα κράτη-μέλη έχουν εγκρίνει εθνικά σχέδια δράσης για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής και ακολούθησαν και τις δικές μας τις συστάσεις. Στο τελευταίο ευρωπαϊκό εξάμεινο, αν θυμάμαι καλά, προτείναμε σε 11 κράτη-μέλη να ενισχύσουν την καταπολέμηση της φορολογικής απάτης και της φοροδιαφυγής και να αναλάβουν τα απαραίτητα εθνικά μέτρα που θα τους επέτρεπαν να βελτιώσουν τη συλλογή των φόρων και επομένως να αυξήσουν τα κρατικά έσοδα στον κρατικό προπολογισμό. Τώρα, όσον αφορά τους στόχους και τους δεσμευτικούς στόχους, στους οποίους αναφερθήκατε. Ενδιαφέρουσα η προσέγγιση αυτή. Να καταφέρουμε δηλαδή να πατάξουμε την λεγόμενη μη δηλωμένη οικονομία. Το πρόβλημα όμως που έχουμε τελικά είναι ότι δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή συγκεκριμένες μετρήσεις του φαινομένου αυτού. Δεν έχει γίνει μία σαφής αξιολόγηση της κατάστασης. Και όταν λείπουν συγκεκριμένα δεδομένα για έναν δεδομένο τομέα, τότε είναι πολύ δύσκολο να καταρτήσει κανείς μια συγκεκριμένη πολιτική, καθώς επίσης και στόχους για την καταπολέμηση του προβλήματος. Είμαι λοιπόν στη διάθεσή σας ε, για την υποβολή προτάσεων από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για το συγκεκριμένο αυτό τομέα και πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το συγκεκριμένο αυτό πρόβλημα. Νομίζω ότι ε, ήδη αναφέρθηκα στο ζήτημα του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου να προσθέσω απλώς ότι ε, στο τρέχον ευρωπαϊκό εξάμεινο θέλουμε να γίνουμε ακόμα πιο σαφείς όσον αφορά τις συστάσεις που απευθύνουμε σε ορισμένα κράτη-μέλη για την καταπολέμηση της ε, φοροδιαφυγής, φοροαποφυγής και φορολογικής απάτης. Θεωρώ λοιπόν ότι ε, το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο αποτελεί ένα ακόμα μέσο, ένα ακόμα εργαλείο που θα μας βοηθήσει να πιέσουμε τα κράτη-μέλη να εφαρμόσουν τις συστάσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το είπατε και η ίδια κυρία Κλέβα ότι ε, οι συστάσεις αυτές δεν είναι δεσμευτικές. Ωστόσο, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου έχουμε προτείνει στα κράτη-μέλη εκείνα τα οποία δεν έχουν εφαρμόσει ακόμα τις συστάσεις μας να το κάνουν ταχύτατα. Κατά αυτόν τον τρόπο θα καταφέρουν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις που απορρέουν από το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο. Ξέρετε ότι ε, οι ειδικέ αναχώρασεις τάσεις το Μάιο του 2014 θα υποβληθούν, βρίσκεται σε εξέλιξη όμως η όλη εργασία αυτή τη στιγμή και η ιδέα την οποία προτείνεται την χάνει επεξεργασία και από μένα και από την ομάδα των συνεργατών μου. ΕΛΚ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, και ζητώ συγγνώμη που έφτασα τόσο αργά, αλλά έπρεπε να παραμείνω στην Επιτροπή των Γυναικών για να ψηφίσω. Έγιναν ηρωικές διαδικαστικές συζητήσεις πρωτού περάσουμε στην ψηφοφορία. Ζητώ συγγνώμη λοιπόν να θέσω ερώτημα για ένα ζήτημα που ήδη έχει συζητηθεί, αλλά με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Επίτροπε, μετά την καταστρεπτική νομική γνωμοδότηση του Συμβουλίου για την πρότασή σας σε ε, σχέση με την ενισχυμένη συνεργασία για τον φόρο επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, πιστεύετε πως ε, η θέσπιση αυτού του φόρου σε αυτό το επίπεδο θα είναι κάτι υλοποιήσιμο όσο ζω τουλάχιστον εγώ ακόμη. Μία μειοψηφία κρατών μελών μπορεί να υποχρεώσει την πλειοψηφία κρατών μελών να υποστούν τις προφανείς επιπτώσεις της ε, θέσπισης ενός φόρου που δεν θέλουν να βλέπουν ούτε ζωγραφιστό για τους γνωστούς σε όλους ε, λόγους. Και ίσως ε, Ε, ε, ίσως, ε, τι να πω, είναι ευαίσθητο το ζήτημα, αλλά οι insiders ε, μου λένε ότι θα μπορούσε να, να πραγματοποιηθεί. Εσείς τι λέτε. Thank you, Mrs. and uh, I ε, απάντησα ήδη σε αυτό το ερώτημα όταν ε, απάντησα ε, στον κύριο Έπινγκ. Αλλά, Σάρων, αν μου το επιτρέψεις να επαναλάβω την απάντηση. Λοιπόν, είπα, από δύο οπτικές γονείς μπορούμε να δούμε το ζήτημα. Ας τονίσουμε πρώτα το τι σημαίνει η νομική γνωμοδότηση του Συμβουλίου. Πρόκειται για με μία συγκεκριμένη παράγραφο ενό συγκεκριμένου άρθρου της πρότασης για τον φόρο χρηματοπιστωτικών συναλλαγών. Η γνωμοδότηση δεν φέρει επί του συνόλου της πρότασης. Θεωρεί η Επιτροπή πως ε, η γνωμοδότηση της νομικής υπηρεσίας του Συμβουλίου είναι εσφαλμένη και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήδη εξέδωσε έκθεση όπου παρουσιάζει ολόκληρη την ε, επιχειρηματολογία ε, που εξηγεί την ε, εγκυρότητα αυτής της παραγράφου και αποδεικνύει ότι συνάδει πλήρως με τις διατάξεις της συνθήκης αυτή η πρόταση Η πρόταση θα παρουσιαστεί στην επόμενη συνεδρία της Ομάδας του Συμβουλίου που θα λάβει χώρα στις 12 Δεκεμβρίου 2013. Το δεύτερο η δεύτερη πτυχή που θέλω να τονίσω είναι ότι τώρα ε, είμαστε στη διαδικασία ενισχυμένη συνεργασία. Αυτό τι σημαίνει. 11 κράτη-μέλη σε εθελούσια βάση και το τονίζω, το τονίζω, ότι ζήτησαν ε, από την Επιτροπή να καταθέσει πρόταση για ένα αρμονισμένο σύστημα φόρου επιχρωματοπιστωτικών συναλλαγών σε αυτά τα 11 κράτη-μέλη. Φυσικά, ο μηχανισμός ενισχυμένης συνεργασίας προβλέπει τη δυνατότητα επέκτασης του πεδίου και συμπερίληψης άλλων κρατών μελών. Προς το παρόν όμως, Αυτά τα 11 κράτη-μέλη θέλουν να προχωρήσουν. Στα χέρια τους είναι τώρα να συμφωνήσουν για το συγκεκριμένο πεδίο εφαρμογή στην αρχιτεκτονική της πρότασης. Και πιστεύω ότι η συμβολή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μέσω της έκθεσης που εγκρίθηκε με πάρα πολύ μεγάλη πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο τροφοδοτεί τη συζήτηση για αυτό το ζήτημα. Τώρα είναι στα χέρια των 11 κρατών μελών να δείξουν πολιτική δέσμευση για να καταλήξουν σε συνένεση και πραγματικά ελπίζω να καταδείξουν ότι έχουν, αναλαμβάνουν αυτή την πολιτική δέσμευση. Αν υποδηματά, τελευταία ερώτηση. Thank you very much. Uh, Ευχαριστώ, Σάρον. Θα μιλήσω στα ελληνικά. And I'll try to combine a little bit the issues that have been uh, raised from my colleagues. Uh, η καταπολέμηση της φορολογικής απάτης, της φοροδιαφυγής, ε, των φορολογικών παραδείσων, γενικότερα η προσπάθεια αποκατάστασης της ε, φορολογικής δικαιοσύνης. Εγώ σε αυτό το πλαίσιο θα εντάξω και αυτό που θέλω να σας ρωτήσω για το φόρο χρηματοπιστωτικών συναλλαγών. Γιατί θεωρώ ότι είναι ένα φορολογικό εργαλείο που εντάσσεται σε αυτή την συνολική προσπάθεια σε όλα τα επίπεδα για αποκατάσταση της φορολογικής δικαιοσύνης. Θέλω να επανέλθω στα ερωτήματα των συναδέλφων Τάισεν και της κυρίας Κλίβα. Γιατί αυτά είναι ζητήματα που ε, δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά στο εθνικό επίπεδο. Ούτε ο φορολογικός ανταγωνισμός, στο πλαίσιο της φορολόγησης των επιχειρήσεων, ούτε η καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής, ιδιαίτερα ε, η φοροδιαφυγή του μεγάλου πλούτου, στο πλαίσιο φορολογικών παραδείσων είτε εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης είτε έναντι τρίτων προορισμών όλα αυτά χρειάζονται ε, δράσεις συγκεκριμένες στο ευρωπαϊκό επίπεδο είπατε μόνο σας αναφερόμενο στην Ελλάδα ότι έχουν γίνει βήματα στη βελτίωση των φορολογικών εσόδων αλλά μένουν ακόμη πολλά να γίνουν. Στο εθνικό επίπεδο όμως είναι περιορισμένα αυτό που μπορούν να γίνουν. Πρέπει να γίνει μια προσπάθεια πιο συστηματική. Αυτό ήταν το μήνυμα και από τον Γενικό Γραμματέα του ΟΣΑ στη συζήτηση που είχαμε πριν. Έτσι. Πρέπει να γίνουν προσπάθειες στο ευρωπαϊκό και σε παγκόσμιο ε, επίπεδο για να μπορέσουμε να προωθήσουμε με αποτελεσματικότητα αυτά τα ζητήματα που είναι κεφαλαιόδου σημασίας. Και σας ρωτώ, ε, είπε η κυρία Κλίβα ότι το Κοινοβούλιο έχει πάρει αυτή την πρωτοβουλία για ένα ψήφισμα με το οποίο θα ζητάει από την Επιτροπή, για να μην παίζουμε τον blame game μεταξύ μας. Τα κράτη-μέλη έχουν ευθύνη. Το Κοινοβούλιο ζητάει από την Επιτροπή όμως να υιοθετήσει αυτή την προσέγγιση για μετρήσιμους συγκεκριμένους στόχους στην, στον περιορισμό της φορολογικής απάτης και στην μείωση της φοροδιαφυγής και έχουμε τώρα το expertise, το know-how γιατί υπάρχουν αυτοί οι μετρήσιμοι στόχοι μέσα για παράδειγμα στα προγράμματα προσαρμογής που εφαρμόζονται στις χώρες με πρόγραμμα, όπως είναι η δική μου. Γιατί λοιπόν σε αυτήν την λογική αυτό, αυτούς τους μετρήσιμους ε, στόχους για τον περιορισμό της φοροδιαφυγής δεν μπορούμε να τους ε, εντάξουμε μέσα στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού ε, Εξαμήνου. Και τελευταία ερώτηση, κύριε Επίτροπε, ε, τι νομίζετε ότι πρέπει να γίνει το επόμενο εξάμεινο και στο πλαίσιο της ελληνικής προεδρίας που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για αυτά τα ζητήματα της καταπολέμησης φοροδιαφυγής για να προωθηθούν, για να υπάρξουν αποτελεσματικές απαντήσεις και στο φόρο χρηματοπιστωτικών συναλλαγών με δεδομένο ότι είναι η πρώτη χώρα από τις 11 που αναλαμβάνει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέλω να σας ρωτήσω ε, ε, εάν περιμένετε να αναγορεύσει σε προτεραιότητα το φάκελο του φόρου χρηματοπιστωτικών συναλλαγών και αν θεωρείτε ότι εξακολουθεί να είναι ρεαλιστικός ο στόχος να κλείσουμε αυτή τη διαπραγμάτευση στο πλαίσιο του τρέχοντος εξαμήνου πριν τις ευρωεκλογέ, όπως έχει ζητήσει κατ' επανάληψη το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ. Well, so, um, λοιπόν, πρώτα απ' όλα να πω πως έχει κομισιόν τώρα, δεν, κατηγορεί κράτη-μέλη. Εάν δείτε τις προτάσεις που κατατέθηκαν στη θητεία αυτή της Κομισιόν, νομίζω τα πει στην ε, η μερίδα που είχαμε για τον ΦΠΑ ήταν η πιο παραγωγική θητεία της Κομισιόν στον τομέα της φορολογίας. Και νομίζω πως ε, σημαντικό είναι το ότι τα κράτη-μέλη ήδη έχουν υιοθετήσει πολλές ε, σημαντικές ε, προτάσεις και ξεκίνησαν τη δουλειά βεβαίω. και άλλα πολλά είναι στο πρόγραμμα ακόμα και ο φόρο χρηματοπιστωτικών συναλλαγών μεταξύ αυτών. Συμφωνώ μαζί σα πω ε, πρέπει να έχουμε και κάποια πολιτική δέσμευση των κρατών μελών που συμμετέχουν για να ολοκληρωθούν αυτές οι διαπραγματεύσεις πριν από τις ευρωεκλογέ. γιατί βεβαίως αυτό είναι σημαντικό και από εθνική σκοπιά. Πολλά, αν όχι όλα τα κράτη-μέλη που αποφάσισαν ε, να συμμετάσχουν στην ενισχυμένη συνεργασία, ε, ε, βλέπουν αυτό το ζήτημα ως ένα σημαντικό πολιτικό ζήτημα στο εθνικό επίπεδο. Χρειάζεται τώρα λοιπόν να εργαστούμε αποτελεσματικά, να εργαστούν δηλαδή τα κράτη-μέλη, να βρουν έναν συμβιβασμό και η Κομισιόν θα κάνει ό,τι μπορεί για να διευκολύνει την εξέβρεση συμβιβασμού. Αλλά βεβαίως ε, επαφίεται στα κράτη-μέλη. Αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορώ να τα εξαναγκάσω εγώ να σηκώσουν το χέρι. Είναι δική τους απόφαση. Όσον αφορά τους δεσμευτικούς στόχους, την καταπολέμηση της ε, φορολογικής απάτης και φοροδιαφυγής. Ενδιαφέρουσα ιδέα. Βεβαίως πρέπει να το δούμε... Ναι, ναι, ναι, ναι έτσι. Ε, να το δούμε πιο στενά. Αν δείτε ιστορικά το ευρωπαϊκό εξάμεινο, κάθε χρονιά περνάει βελτιώνουμε το πεδίο εφαρμογή ε, τους στόχους ε, των συστάσεων και είναι κάτι το οποίο εξελίσσεται. Θα έχουμε, τέσσερις, ε, θα έχουμε τέταρτο γύρο ευρωπαϊκού εξαμήνου και είναι κάτι το οποίο αναλύεται και εντός του Κοινοβουλίου και οι ιδέες που ακούγονται θα μπορούσαν να συνεισφέρουν σε ολόκληρη την διαδικασία του ευρωπαϊκού εξαμήνου και χαίρομαι ιδιαίτερα για το ότι η φορολογία είναι αναπόσπαστο τμήμα της ε, διαδικασίας και μπορούμε να κάνουμε πολλά πρακτικά πράγματα στο πεδίο του συντονισμού της φορολογίας που πιθανώς δεν θα μπορούσαν να αποτελέσουν ευρωπαϊκή νομοθεσία λόγω περιορισμών επικουρικότητας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Επίτροπε. Πράγματι θα μου τη θυμίζετε συνεχώς αυτή την, την ε, παρατηρήσή μου, αλλά είναι αλήθεια. Είδα ότι το, το γράψατε και στο Twitter. Αλλά όπως είπα ισχύει, είναι αλήθεια. Και όπως ξέρετε προσπαθούμε να κάνουμε κάποια πράγματα καινοτόμα στον τομέα της φορολογίας με τη δημοσίευση μη οικονομικών πληροφοριών γιατί θεωρούν πως η δημοσίευση είναι ένας μηχανισμός που μπορεί να βοηθήσει στο να λειτουργεί η φορολογική βάση κτλ. Οπότε αν το επιτύχουμε βεβαίως θα οφείλεται σε εσά και στον ΩΣΑ τον οποίο κλέψαμε ιδέες. έστω και αν τελικά δεν ε, θα πιστωθεί σε εσά. Νομίζω λοιπόν πως η πλειοψηφία της Επιτροπής μας είναι υπέρ της επιτυχίας αυτής, αν και θα πρέπει νομίζω να πιέσουμε την Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων και τα κράτη-μέλη σε πολλά από αυτά τα ζητήματα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αναμένουμε την επόμενη συνάντησή μας. Όποτε την κανονίσουμε. Σας ευχαριστώ. Συνάδελφοι, θα ξεκινήσουμε αργότερα το απόγευμα, 3 και 45. Παρακαλώ να είστε στην ώρα σας γιατί θα ξεκινήσουμε αμέσως με τις ψηφοφορίες. Αν δεν υπάρχουν αρκετοί και βγουν περίεργα τα αποτελέσματα δεν θα φταίω εγώ.